του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012, ως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, καθώ και έκθεση του κ. Μπέγκερ για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξία. Πηγαίνουμε λοιπόν στη συζήτηση. Η συνάδελφό μα, η Φρανσέσκα Μπαλτζάνη, θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Είναι η συγγήτρια όσον αφορά αυτή την έκθεση. Κυρία Μπαλτζάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζούμε στιγμές κρίσης και αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και είναι κρίση εμπιστοσύνη. Κρίση εμπιστοσύνη που πλήττει όλους τους ε, πολίτες, κυρίως τους ε, νεότερους που έχουν περισσότερες δυσκολίες να έχουν το θάρρος και τη βούληση να οικοδομήσουν το μέλλον τους. Για να καταπολεμηθεί αυτή η κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια πρόκληση, με πρόκληση απέναντι τη που έθεσε, τη μεγάλη στρατηγική για το 2020, για την Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική που θα πρέπει πάντα να αντισταθεί σε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη. Να μας οδηγήσει σε ένα μονοπάτι προς ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερο επίπεδο ζωής. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε στο επίκεντρο του προπολογισμού του 2012 τη χρηματοδότηση αυτής της στρατηγικής ξεκινώντας από την πρώτη από τις προτεραιότητες. Μια Ευρώπη με καλύτερη απασχόληση, περισσότερη απασχόληση, με ποιοτική απασχόληση. Μια Ευρώπη που βασίζεται στην καινοτομία, στην έρευνα. Και γι' αυτό σαν κοινοβούλιο ζητήσαμε και ζητούμε περισσότερους πόρους για τα προγράμματα κλειδιά. Τα τρία, τους πραγματικούς κινητήρες της στρατηγικής του 2020. Το πρόγραμμα Lifelong Learning, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα CHIP Πρέπει να έχουμε συνοχή λοιπόν, συνεπείς να δώσουμε συνέχεια στις προθέσεις μας, ε, να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, συνεπώς, τη συγκεκριμένη ε, κατασκευή αυτής της διαδρομής. Να μην χρηματοδοτήσουμε μία στρατηγική... εάν κατασκευάσουμε μια ε, πολιτική για την κρίση αυτή τη στιγμή, να μην τη χρησιμοποιήσουμε τώρα που είναι η κρίση, θα ήταν κακό μήνυμα. Περιμένουν σοβαρότητα και συνοχή πολίτε και αγορέ αγορές. Ε, ιδιαίτερα προσέχουν τις αποφάσεις που παίρνουμε, τη δυνατότητά μας ε, εγκαίρως να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερο ευαίσθητο, ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα να δώσουμε θετικά μήνυματα. Προ αυτή την κατεύθυνση θα ήταν έξοχο να έχουμε ένα προπολογισμό πραγματικά αρχίζει να δρομολογεί τη θετική του 2020, αλλά θα ήταν σημαντικό να το κάνουμε αυτό ε, μέσω μεγάλη θεσμική συνεργασία για να στείλουμε ένα καλό μήνυμα ότι αυτό το κοινοβούλιο θεώρησε ότι πρέπει να δώσει μεγάλη αξιοπιστία στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιτροπή μας εργάζεται αυτή τη στιγμή των δυσκολίων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό θεώρησε ότι είναι εφικτές οι εκτίμησεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανάγκες των πληρωμών. Υπάρχει και άλλο επίγον θέμα. Ε, στη Μεσόγειο πολλές χώρες αλλάζουν το θεσμικό τους καθεστώς και δεν μπορεί να μείνει η Ευρώπη εκτός αυτού του πλαισίου, δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο του όλου σκηνικού, θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή πολιτική. Άρα υπάρχει ανάγκη να αντιδράσουμε στην κρίση να έχουμε ανανεωμένη ηγετική θέση όσον αφορά το διεθνές προσκήνιο. Για αυτούς τους δύο θεμελιώδεις στόχους ζητούμε να χρησιμοποιηθεί το μέσο ευελιξίας. Και θα είναι σημαντικό, συνεπώς, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε και νικήσουμε αυτές τις προκλήσεις, να δώσουμε εμπιστοσύνη, να δείξουμε ότι υπάρχει αξιοπιστία, να δείξουμε ότι προσέχουμε αυτά τα θέματα και να το δείξουμε στους πολίτες και στους άλλους θεσμούς που κοιτάνε προς τα δώ. Αλλά υπάρχει και άλλη πρόκληση πέραν αυτής τη προκλήσεως. Να καταφέρουμε τα αυτά με διαφάνεια και δεν θέλουμε για τον προπολογισμό να ακολουθήσουμε διαπραγματευτική τακτική. Να δείξουμε ότι θεωρείται θεμελιώδη ο προπολογισμό το 2012. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε σε μια θέση και κοινή σε συγκεκριμένους χρόνους γρήγορα να συμφωνήσουμε για να δώσουμε την εικόνα ότι η Ευρώπη μπορεί ε, να βρίσκει τη θέση της στη σωστή στιγμή. Να στέκεται στα πόδια της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαλζάνη. Επόμενος ε, αγορητής, ο Ζωζέν Μανουέλ Φερνάντες, που επίσης είναι εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία περίοδο χρηματοπιστωτικής αλλά και κοινωνικής ε, κρίσης και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μία ιδιαίτερη προσπάθεια όλα τα θεσμικά όργανα μαζί και θα πρέπει να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η στιγμή που διανύουμε είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους έχουν καταλάβει τα άκρα είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά στους εξτρεμιτιστές να παρουσιάσουν δημαγωγικό, δημαγωγική σκέψη η οποία θα τους επιτρέψει επιτρέψει να προωθήσει τις δικές τους ακραίες ε, και εθνικιστικές θέσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να ε, αφήσουμε στην άκρη τις προσπάθειες που έχουν κάνει όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρουσιάσουν αυτό τον προϋπολογισμό. Βλέπουμε λοιπόν πως η τα διοικητικά έξοδα φτάνουν μόνο στο 5,59% ε, του συνολικού προϋπολογισμού. Ε, βλέπετε λοιπόν πως έχουμε ήδη ξεπεράσει τα όσα μας είχαν ζητηθεί ε, γιατί η εξοικονόμηση που έχουμε στον τομέα 5 είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έχουμε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις. Όμως Έχουμε και πάρα πολλέ δαπάνε οι οποίες θα προβλέψουμε, γιατί ενδέχεται η Κροατία να γίνει μέλος μας και επίσης έχουμε και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πως το 2012 ε, έχουμε ε, καταφέρει μια αύξηση τη τάξη του 1% που είναι αρκετά χαμηλότερη από την, την αριθμική αναπροσαρμογή που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει. θα ήθελα να στραφώ προ το Συμβούλιο, αλλά ε, απευθυνόμενοι στο Συμβούλιο, θα ήθελα να τους ζητήσω ε, να καταλάβουν πως έχουμε κάνει ε, μεγάλη προσπάθεια για να μειώσουμε τις διοικητικές μας δαπάνες ε, και βρισκόμαστε στα όρια των όσων μπορούμε να αντέξουμε. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες ε, είμαστε υποχρεωμένοι να καλύπτουμε. Εξόδα συντήρησης, λογαριασμού ηλεκτρικού. Δεν μπορούμε να μην τις πληρώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προσπάθειες που έκαναν οι πολιτικές ομάδες και το Προεδρείο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία και σε πραγματική οικονομία διαστρωτική. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσει σε επίπεδο ε, Προεδρείου καταφέραμε να μειώσουμε κατά 74 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ τις απαιτήσει που είχαμε για παράδειγμα σε συνεδριάσεις συνδιαλλαγής. Για το 2012 είπαμε πως θα έχουμε το χαμηλότερο ρυθμό ε, τέτοιων συνεδριάσεων ε, ιστορικά ε, για την Κροατία και εκεί έχουμε κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Το Συμβούλιο κατάφερε να μας εντάξει ένα ποσό. Έχουμε μια επικαιροποίηση του 1,9% που είναι και αυτό κάτω από την αύξηση του πληθωρισμού για να καλύψουμε και την είσοδο της Κροατίας αλλά καταλαβαίνετε πως τα όσα ε, κάναμε τον ε, Απρίλιο ε, δεν φτάνουν για να καλύψουν τα 18 νέα μέλη που έχουμε και το θέμα της Κροατίας. αν συγκρίνουμε με το 2011, γιατί μιλάμε και για μια περαιτέρω μείωση 25,1 εκατομμύριο ευρώ, θα δείτε πως έχουμε δύο, δύο μεγάλες δαπάνες. Έχουμε την Κροατία και το 18 νέα μέλη του Κοινοβουλίου μας που μας οδηγούν σε μια αναγκαστική επικαιροποίηση ε, του προπολογισμού μας. Παρόλα αυτά η αύξηση είναι η χαμηλότερη που έχουμε προτείνει ποτέ. Εμείς λοιπόν θα διατηρηθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πρόοδο έτσι ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να καλύψουμε τα όσα ζητούν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο συνάδελφος ε, Ράιμερ Μπέργκε, ο εισηγητή, έχει το λόγο επίσης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Βρισκόμαστε στη βάση του άρθρου 27 της Συμφωνίας ε, της Διαθεσμικής, ε, της Εργονικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σε ό,τι αφορά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Θα ήθελα να πω όμως στη συζήτηση επίσης ότι η έκθεση αυτή, η οποία ψηφίστηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, δεν θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, γιατί Είμαστε πιστοί στην σύμβαση. Ξέρουμε ότι το μέσο της ευελιξίας ε, μπορεί να, κινηθεί, να κινητοποιηθεί μόνο από κοινού από τι δημοσιονομικέ αρχέ, αλλά θεωρούμε ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη σε ό,τι αφορά την στρατηγική του Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, σε ό,τι αφορά την κατηγορία 1α, να τη στηρίξουμε με 30,75 εκατομμύρια και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, να τη στηρίξουμε με επιπλέον 208 1,67 εκατομμύρια ευρώ λόγω των εξελίξεων στην ε, γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δέσμευσή του για έναν ε, καλό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν ε, του αξίζει στην κοινή γνώμη και στον τύπο να του ασκείται κριτική από το Συμβούλιο. Κοιτώντας τις δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή ε, Προπολογισμού βρίσκονται λίγο πιο πάνω από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Αλλά υπάρχουν εδώ κάποιες κλασικές διαφορές. Το Συμβούλιο ή τμήματα του Συμβουλίου εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός αποτελεί ένα εχθρικό στοιχείο και ξεχνούν ένα πράγμα, αμελούν μία διάσταση ότι οι δεσμεύσει οι οποίες έχουν αναλυφθεί κάποια στιγμή θα πρέπει να μετατραπούν σε πληρωμές και όσο πιο καθυστερούμε τόσο πιο μεγάλη θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη τελική ανάλυση. Και αυτό λοιπόν είναι το θέμα όταν ε, καταρτίζουμε την δημοσιονομική πολιτική και θα πρέπει να πούμε στην κοινή γνώμη ότι μεταξύ του 2000 και του 2010 οι εθνικοί προϋπολογισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 62% ενώ ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο κατά 7% και παράλληλα με αυτή την αύξηση χρηματοδοτήθηκε και η διεύρυνση. Το 11. πολλά κράτη-μέλη ξοδεύουν παραπάνω 23% κατά μέσο όρο τα κράτη-μέλη από το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό θα είναι 24% το επόμενο έτος και θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που θα ψηφίσουμε σήμερα αποτελεί μια πολύ σόφρον πρόταση για τον προϋπολογισμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που ήταν εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταφέραμε να καταρτήσουμε έναν προπολογισμό με μία αύξηση μόνο 0,8% χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη Λισαβόνα και την ε, Κροατία. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό κυρίε και κύριοι να τονίσω ότι στην κατάσταση αυτή όπου κάναμε τα μαθήματά μας για τον προπολογισμό για το έτος αυτό δεν έχει νόημα τα επόμενα χρόνια θα πρέπει όλοι οι θεσμοί, όλα τα θεσμικά όργανα να σκεφτούν πού μπορούν να μειωθούν τα έξοδα σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία σε όλα τα θεσμικά όργανα χωρίς να παρεμποδιστεί η λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πακέτο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο και θα πρέπει να συμβάλλει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι για τις ε, παρεμβάσεις σας και τώρα εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ο κύριος Υπουργός. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άκουσα με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Καλωσορίζω τη εκφράση μετάφραση αυτή της πρόθεσης να θετηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για τον προπολογισμό του 2020 καταβάλλονται προσπάθειες φοβερές στα διάφορα κράτη-μέλη και δέχονται πιέσεις. Επουδενή δεν θέλουμε να στείλουμε αρνητικά μηνύματα προς τον κόσμο τη στιγμή που τα κράτη-μέλη προσπαθούν να εξηγιάνουν τα οικονομικά τους. Τα κράτη-μέλη έχουν πετύχει μία συμφωνία με μικρή διαφορά ψήφων όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Η αύξηση του 2,9% στην ανάληψη υποχρεώσεων με το 2011, καθώς και το 2,02% αύξηση στις πληρωμές, είναι αυτό που απετέλεσε το αντικείμενο της συμφωνίας. Το Συμβούλιο προσπάθησε να μην ξεπεράσει τα ανώτατα όρια της πολιετούς ε, οικονομικής ε, περίοδου, δημοσιονομικής περίοδου. Το Συμβούλιο θέλει να είναι έτοιμο και σε θέση να εξασφαλίσει ότι παραμένουν τα αποθεματικά για κάποιες απρόβλεπτες ε, περιστάσεις μας ανησυχούν κάποιες τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ξεπερνούν τα ωρία το Συμβούλιο ανησυχεί για κάποιες ψηφοφορίες που ε, επέρχονται στον αφορά τις πληρωμές που κάποιες πληρωμές ξεπερνούν και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012. Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να πετύχει τις προτεραιότητες που έχει θέσει, το επίπεδο των πληρωμών όμως θα πρέπει να είναι αρκετό αλλά όχι υπερβολικό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι υπερβολικά επίπεδα πληρωμών οδηγούν σε υπερβολικά ελλείμματα στα κράτη-μέλη. Και απαιτείται δανεισμός. Δοθήσεις της καταστάσεως της, των κεφαλαγορών, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του παρελθόντος και να είμαστε ψύχρεμοι όσον αφορά τον προπολογισμό του 2012. Ανησυχεί το Συμβούλιο για τα σχέδια του Κοινοβουλίου να ψηφίσει αυξήσεις που ξεπερνούν το ανώτατο την οροφή, στην 1α και στο κεφάλαιο 4 κατά 240 εκατομμύρια ευρώ. Στο ύψος αυτό. Όσον αφορά το πρόγραμμα ITER, το Συμβούλιο θα ήθελε να επιτευχθεί ε, σύντομα μια συμφωνία για συμπληρωματική χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Εκφράζει τη λύπη του όμως το Συμβούλιο για την απόρριψη από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της αναμαδοποίησεως τη χρηματοδότηση με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υποστηριχθεί το πρόγραμμα ITER. Ανησυχεί επίση το Συμβούλιο για τα όσα συμβαίνουν και στο κεφάλαιο 1β, όπου το Κοινοβούλιο επιδιώκει αύξηση του 8%. Το Συμβούλιο σημειώνει επίσης τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να περιορίσει την αύξηση στο κεφάλαιο 4 ανησυχεί το Συμβούλιο όσον αφορά τους περιορισμούς που θέτει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πολιτική. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5, το τίτλο 5, ε, το Συμβούλιο θέλει αυστηρούς ελεγχούς περιορισμούς των διοικητικών δαπανών μέσω εντατικής διοργανικής συνεργασίας και αυξημένης αποδοτικότητας, ούτως ώστε οι περιορισμένοι πόροι να ξοδεύονται σωστά στα πλαίσια της γενικής ε, οικονομικής εξυγίανσης που προσπαθούν να πετύχουν και τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πρέπει να υποστηριχθούν μέσω του προϋπολογισμού του 2012. Όμως η διαφορά μας αφορά τα επίπεδα της αναγκαίας χρηματοδότησης. Το επίπεδο κυρίως των πληρωμών θα πρέπει να είναι τέτοιο τόσο ώστε να μην επιβαρύνει υπερβολικά του προπολογισμού των κρατών μελών και να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να περιορίσουν άλλε σημαντικέ δαπάνε που χρηματοδοτούνται από του προπολογισμού των κρατών μελών. Εν κατακλείδη, να επαναλάβω τι ελπίδε και επιθυμίες του Συμβουλίου τα επόμενα στάδια της ε, διαδικασίας του προπολογισμού να ακολουθηθούν επικοδομητικά σε επικοδομητική ατμόσφαιρα, τόσο ώστε όλες οι πλευρές να ικανοποιηθούν με τα αποτελέσματα του προβλησμού του 2012. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Γιάννους Λεβαντόσκη εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη. Στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου συζητήσαμε το κείμενο ε, όπως ε, το κείμενο του Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή συζητάμε λοιπόν το κείμενο του Κοινοβουλίου λίγες ώρες πριν αυτό λάβει την τελική του μορφή. Είναι προφανές πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από το Συμβούλιο για διάφορα και πολύ σημαντικά θέματα. Εάν λοιπόν ε, το Συμβούλιο επιβεβαιώσει τη θέση του που είναι πάρα πολύ πιθανό παρόλο που βρισκόμαστε σε μία ε, εξαιρετικά δύσκολη στιγμή ε, και πρέπει να σου πω ότι βεβαίως είμαστε και οι τρεις εδώ εκπροσωπούμε τρία διαφορετικά όργανα και είμαστε από την ίδια χώρα αλλά νομίζω ότι για τις 21 μέρες που μένουν ε, για να αποφασίσουμε οι θέσεις μας δεν θα αλλάξουν σημαντικά. θα ήθελα τώρα να στραφώ προς τον κύριο Μπόκερ, τον κύριο Φερνάντες και την κυρία Μπαλζάνη. Καταρχήν για το σχέδιο προϋπολογισμού ε, πιστεύουμε πως ε, το Κοινοβούλιο έχει στον τομέα 1α εξαντλήσει τα περιθώρια που υπάρχουν και όχι μόνο έχει εξαντλήσει τα περιθώρια αλλά στο 1α έχει ζητήσει περισσότερο από όσα απαιτούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέσο ευελιξίας. Οι προτεραιότητε που έχουμε βεβαίω μας βρίσκουν σύμφωνο. βρίσκουν σύμφωνο με τον τρόπο που του στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως οι δημοσιονομικοί στόχοι της ε, στρατηγικής για το 2020 που έχουν σκοπό να αυξήσουν θέσει εργασίες θα πρέπει κάπως να συγκεραστούν με τα όσα έχουμε γιατί βέβαια ζούμε σε ένα ε, περιβάλλον δημοσιονομικής στενότητας. Τώρα, για την εξωτερική δράση, εμεί είμαστε υπέρ του μέσου ευελιξία, αλλά ο λόγο που το στηρίζουμε είναι γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική γειτονία. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο. Είναι σημαντικό για όλα τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να επενδύσουμε στη σταθερότητα της γειτονιάς μας. Δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε ε, μόνο με αναδίπλωση από άλλα μέτωπα. Τώρα μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό νομίζω έχει συμφωνηθεί από τα ε, θεσμικά όργανα. Αλλά Νομίζω πως ε, τα όσα προτείνεται για μια απλή αναδίπλωση και νέα χρήση πόρων δεν μπορεί να γίνει. Για το ίτερ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να ε, φεύρει ακόμα μια τροπολογία συμβιβαστική ε, μετά από τις υπόλοιπες που έχει υποβάλει ε, θα λειτουργήσει μόνο αν δείξουμε όλοι καλή πρόθεση. Δεν θα πρέπει να γίνει καυτό θέμα το ίτερ ε, και δεν θα πρέπει να μας σταματήσει αυτό ή να δυσκολέψει τη συμφωνία για τον ε, προπολογισμό του 12. Τώρα για το επίπεδο πληρωμών αυτό πάντα είναι ένα θέμα ευαίσθητο. Στο σχέδιο δικού μας, το δικό μας σχέδιο προπολογισμού είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα παραδώσουν τα 27 κράτη-μέλη και είπαμε επίπεδο πληρωμών θα είναι 9 δις ευρώ κάτω από το περιθώριο που έχουμε για το 2012 γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια αυτό περιορισμού. Λοιπόν, ε, θα σας επιβεβαιώσω πως αυτή τη στιγμή έχουμε μια κινητικότητα στο θέμα των πληρωμών. Συνήθως το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών αυτό γίνεται γιατί φτάνουν πολλά αιτήματα πληρωμών ε, ε, φέτος ε, δεν μιλάμε για πλεονασματικές, για επιπλέον πληρωμές για το 2011, μιλάμε για μείωση πληρωμών για το 2011 και αυτό φαίνεται και από την διόρθωση που έγινε στον προϋπολογισμό. Για την απογραφή λοιπόν των πληρωμών πρέπει να σας πω πως τη θέση που έχουμε για τον περιορισμό των πληρωμών μέσα στα πλαίσια της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, κοιτάξτε, και στην έρευνα και στην τεχνολογία και στην κοινοτομία έχουμε ε, πρόβλημα κονδυλίων για το 2011. Για το διοικητικό προϋπολογισμό, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβετε είναι πως το μεγαλύτερο όργανο που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παγώσει ε, στο ονομαστικό επίπεδο και δεν ζητά άλλες θέσεις. Ξέρουμε όμως πως πάντα ζήτησε ε, απόθεμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή είναι και η πάγια τακτική του, ελπίζοντας πως αυτές οι θέσεις ε, θα απελευθερωθούν. Νομίζω πως ε, είναι γνωστή η θέση μας για τα πειραματικά σχέδια και για τις προετοιμαστικές δράσεις. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τώρα, για την επόμενη πρωτοβουλία που κάναμε, ε, προσπαθήσαμε να απελευθερώσουμε ορισμένα κονδύλια αλλά δυστυχώ, στο Συμβούλιο Γεωργία Περισσότερης της περασμένης εβδομάδα δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο για το καθεστώ αυτό που θα χρηματοδοτεί απόρου και ε, ένα κομμάτι ε, των πληρωμών, 340 ευρώ, μπήκαν στο αποθεματικό από τα 500 που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι εκεί έχουμε χρόνο να δράσουμε για αυτό το σχέδιο έτσι ώστε να απελευθερώσουμε όλο το ποσό για τη στήριξη των απόρων. Πριν τη συνδιαλλαγή, στόχος μας είναι να υποβάλουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εξελίξεις που τρέχουν φέτος στις πληρωμές και όπως πάντα εμείς θα είμαστε ο τίμιος μεσίτης, ο τίμιος διαμεσολαβητής στην προσπάθεια εξέβρεσης ε, ε, συμβιβασμού για το 2012. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, Και τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η κυρία Μαρία Μουνίστερ Κίζα. Ευχαριστώ πολύ. στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και στον εκπρόσωπο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πούμε πως ε, για τον τομέα 4 και πάλι έχουμε υποχρηματοδότηση που δεν θα μας επιτρέψει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης. Εμείς έχουμε θέσει ένα στόχο. Είπαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει παγκόσμιος παίκτη. Με τι πόρους, με πόρους που φθήνουν και πάλι φέτος και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε με τον τομέα 4, η οποία υποχρηματοδοτείται, τι υποχρεώσει που αναλάβαμε στο παρελθόν, που αποτελούσαν πολιτικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαιτούν συνέχεια. Όπω επίση και τι νέε προτεραιότητε, για παράδειγμα, χρηματοδότηση τη Αραβική Άνοιξη, θέμα που προέκυψε φέτο. Στην Επιτροπή λοιπόν Εξωτερικών Θεμάτων φανήκαμε υπεύθυνοι και περιοριστήκαμε όσο μπορούσαμε, έτσι ώστε να καλύψουμε του στόχου που έχουμε και τι προκλήσει. Λοιπόν, θέλουμε να είναι η χρηματοδότηση ε, αυτή που έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Παλαιστίνη, για το μέσο σταθερότητας και λυπάμαι ιδιαίτερα. Λυπάμαι κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος, λυπάμαι κυρία μου, για τα... αλλά δυστυχώς δεν έχετε χρόνο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Επόμενος είναι ο κύριος Γκέρεντς για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, στη γνωμοδότησή τη για τον προπολογισμό του 2012, η Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί τι προτεραιότητε. Καταρχά, στο κατηγορία 4 του προπολογισμού που υποχρεωματοποιείται συνεχώ, εκεί θα πρέπει να γίνουν διορθώσει για να επιτευχθούν οι στόχοι τη χιλιετία για την ανάπτυξη και να υπάρχουν λιγότερε απογοητεύσει. Δεύτερον, η αραβική άνοιξη μα δημιουργεί προκλήσει και δημοσιονομικά Λοιπόν, ε, και δεν, δεν πρέπει να κάνουμε περικοπέ από αλλού, πρέπει να κινητοποιήσουμε συμπληρωματικού πόρου. Το ίδιο ισχύει και η χρηματοδότηση των πολιτικών που θέλουν να μειώσουν τι συνέπειε αλλαγή του κλίματο στι αναπτυσσόμενε χώρε. Μετά θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί όσον αφορά την κατανομή των πόρων μα, να έχουμε καλύτερου στόχου, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στι φτωχέ χώρε και στι πλούσιε και αναδυόμενε χώρε. Οι πλούσιε και αναδυόμενε χώρε δημιουργούν επαρκεί πόρου για να ε, μειώσουν τη φτώχεια εντό των συνόρων. Και μετά Πιστεύουμε τέταρτον ότι χωρί καινοτόμε χρηματοδοτήσει, κυρίω και χωρί την φορολόγηση των χρηματοδοτικών συναλλαγών, θα μα λείψουν τα μέσα για να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου που καθορίσαμε οι ίδιοι στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Συνένεση στην Ανάπτυξη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Πέτερ Σνάσνη τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε καιρού οικονομικών προβλημάτων και δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να εξακολουθήσουμε τι επενδύσει. Θα στραφούμε στην ε, ανάπτυξη και στην ευημερία του αύριο. Στην Επιτροπή Ιστορικού ε, διεθνού Εμπορίου έχουμε εγκρίνει τέτοιε πρωτοβουλίες μια πλατφόρμα συντονισμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή στο παγκόσμιο ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα αποτελούν δύο προτάσεις οι οποίες πέρασαν από την Επιτροπή μας σχεδόν ομόφωνα. Η πρώτη ανοίγει την πόρτα σε πολύ πιο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στην ε, διεθνή ανάπτυξη και η δεύτερη πρωτοβουλία σκοπεύει, αποσκοπεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βόρεια Αφρική. Τα μέλη της Επιτροπής μου ε, διέκριναν τα σαφή ωφέλη των ε, πρωτοβουλειών αυτών και ελπίζω ειλικρινά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο Λε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το βασικό μήνυμα της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων είναι ότι θα πρέπει οι νέες εποπτικές αρχές να λάβουν τους πόρους που χρειάζονται για να μπορούν να επιτελούν το έργο τους. Είναι καλό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αποστέλει ένα μήνυμα προκειμένου να λάβουν όντω τα μέσα που χρειάζεται για να ανταποκριθούν στην εντολή τους αυτές οι νέες υποπτικές αρχές. Ευρωπαϊκή εποπτική, ε, ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος των Τραπεζών και το stress test μας κατέδειξε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος. Ε, κατέδειξαν τα stress test του Ιουλίου ότι τα εθνικά συμφέροντα και τα λόμπι κυριαρχούν σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά τους. Τώρα θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν ο έλεγχος, αλλά δεν έχουμε μια σωστή εικόνα για το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Θα πρέπει στο επόμενο τεστ να είναι ανεξάρτητες εντελώ οι εποπτικές αρχές και γι' αυτό χρειάζονται λοιπόν οι απαραίτητοι πόροι. Κυρία Περβάνης Περές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά την, την υποστήριξη του σχεδίου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα κονδύλια που αφορούν την Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίτροπο ήθελε να το υποστηρίξει, θέλαμε να το τονίσουμε και εμεί. Αυτό ο προπολογισμό από 14 Ιανουαρίου ενιστότο έτου είναι ο πρώτο προπολογισμό μετά την δημοκρατική επανάσταση στις αραβικές χώρες και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την κατάρτιση το χαιρετίζουμε που δημιουργήθηκε για το κοινωνικό διάλογο, για την ανάπτυξη αγορά εργασία, για το διάλογο που θέλουμε να κάνουμε με αυτούς τους εταίρους των νοτίων ακτών της Μεσογείου ε, να μπορέσουν όλοι αυτοί να υποστηριχθούν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δυστυχώ αυτό ο προπολογισμό δεν είναι ο πρώτο τη περίοδου κρίσεω που αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, όλη η δράση που θα μπορούσε να αναλυφθεί για την υποστήριξη απασχόληση των νέων, κυρίω μέσω των πιλωτικών προγραμμάτων που δρομολογήσαμε και με το πρόγραμμα τη πρώτη δουλειά για του νέου, τι πρώτε θέσει απασχόληση για του νέου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στη συναλλαγή του προπολογισμού να παραμείνουν αυτά τα κονδύλια εντό του πλαισίου που ψηφίσαμε. Ευχαριστώ. κυρία Γιούτα Χάουγκ έχει το λόγο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην υποκρινόμαστε γιατί στη διαδικασία του προπολογισμού ε, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε κάθε χρόνο. Μπροστά σε ένα συμβούλιο που δεν μας καταλαβαίνει. Το συμβούλιο πάντα περικόπτει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και στη, μικρό αυτό, στη μικρή αυτή χρηματοδότηση για θέματα ε, κλίματος και περιβάλλοντος μαζί με όλες τις υπηρεσίες ούτε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για 0,67% ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Γι' αυτό χαιρόμαστε που η Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, επανησύγα για τις προτάσεις της Επιτροπής μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Φραντσέσκα Μπαλτζάνη, την εισηγήτρια, η οποία έκανε εξαιρετικό έργο. Επίσης χαιρόμαστε που το πακέτο το οποίο προτάθηκε προτείνει 7 πλητικά προγράμματα και τρία μέτρα προετοιμασίας. Ποτέ δεν είχαμε πετύχει μια τέτοια επιτυχία. Τώρα ίσως θα μπορούσαμε για μία φορά στις διαπραγματεύσεις από κοινού με το Συμβούλιο να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Ράινχαρτ Μπιουτικόφα από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Βιομηχανίας ήταν κοινή υπεποίθηση από όλε τι πλευρέ ότι οι προτεραιότητε του προπολογισμού θα πρέπει να αποτυπώνουν του στρατηγικού στόχου τη Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγικής το 2020 και χαιρόμαστε που μα υποστήριξε στη θέση μα η Επιτροπή προπολογισμού Στην Επιτροπή μα. είχαμε τρει βασικέ προτεραιότητε. Καταρχά η ανάγκη του FP7 να χρηματοδοτηθεί για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και να βοηθήσει στην ανταπόκριση στις ε, προκλήσεις. Δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν χρήματα από το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7 πρόγραμμα πλαίσιο. Ξέρουμε ότι θα είναι ε, μεγάλη η μάχη που θα δοθεί με το Συμβούλιο. Κατά δεύτερον, στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν αποδεχθεί χρήσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τρίτον, θα πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες στην ενεργειακή πολιτική και χαιρόμαστε που η Επιτροπή Προϋπολογισμού μας υποστήριξε στις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ και τώρα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ ο συνάδελφος Έντουαρτ Κοζούνσνικ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Όλοι τώρα συζητάνε για το θέμα της κρίσης. Πραγματικά ζούμε σε συνθήκες κρίσης και κάνουν τεράστιες περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα ήταν τελείως ακατάλληλο να έχουμε αύξηση πάνω από το 2% στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 4,9% που προτείνεται εμένα μου δημιουργεί την εντύπωση πως οι συντάκτες του προϋπολογισμού ε, ζουν σε ένα κόσμο ουτοπικό και φανταστικό. Εγώ είμαι υπέρ βεβαίως προϋπολογισμού ανάπτυξης, αλλά αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας κανείς ένα διαφορετικό φιλοσοφικό δόγμα. Δεν χρειάζονται οριζόντιες αυξήσεις. Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος απόδοσης των έργων και όσα δεν είναι βιώσιμα και δεν λειτουργούν θα πρέπει να εγκαταληφθούν και να ε, στοχεύσουμε τις ε, προσπάθειές μας ε, και τα κονδύλια στην εσωτερική αγορά που θα εξασφαλίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε στον κύριο Λιβεράτσκι το λόγο που είναι στην Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού. Επιτροπέ, Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα έπρεπε να αποτελέσουν τη δική μας προτεραιότητα, πιστεύω. Τουλάχιστον είναι η προτεραιότητα της δικής μας Επιτροπής. Και η πρόταση που έγινε για μία μείωση της τάξης του 10% στον ε, τομέα αυτό νομίζω ήταν η μεγαλύτερη που προτάθηκε για οποιοδήποτε τομέα. Ε, για μας το θέμα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Τα κράτη-μέλη θεωρούν πως τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα ε, βοηθήσουν και νομίζω ότι αποτελούν προτεραιότητα και για εμάς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέρη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να κατανοήσω τα λεγόμενα του κύριου Υπουργού γιατί μας είπε πως οι πληρωμές δεν θα πρέπει ε, να έρθουν σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες και θα πρέπει να συνδυάζονται. Άρα λοιπόν ο Επίτροπος κύριος Λεβαντόφσκι ο οποίος θέλει να ε, γίνει ε, τίμιος ε, διαμεσολαβητής θα έπρεπε να εξασφαλίσει πως αυτό θα συμβεί. Περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κύριος Λάσλο Σούριαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλωσόρισε τις αποφάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών ζητούμε από το Κοινοβούλιο να μην αλλάξει την ουσία των όσων αποφασίστηκαν. Συμφωνούμε μεταξύ μας και η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα, λαμβάνει η χώρα με το Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις πληρωμές για αναπτυξιακή βοήθεια, για αυτό το θέμα θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ε, να υπάρχει καθυστέρηση όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια Μιλήσαμε για περικοπές 9 δισεκατομμυρίων, αλλά στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν μπήκαμε στη συζήτηση, δεν θέλαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις και παζάρια. Θεωρήσαμε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνδιαλλαγή θα χρειαστεί να υπάρξει ένα συμβιβασμός και απαιτείται πολιτική βούληση από πλευρά των Υπουργών που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων. Ο κ. Κάπουλα Σάντο, στην Επιτροπή Γεωργία. Ε, Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, ε Πολωνική Προεδρία. Ο γεωργικός ε, κλάδος ε, στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη για να έχουμε καλής ποιότητας ε, τρόφιμα που θα εξασφαλίζονται στους καταναλωτές σε καλές τιμές με ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι βιώσιμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα προϋπολογισμό γεωργικό ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες μας για το 2012. Θα ήθελα να σας υπογραμμίσω και να συγχαρώ βέβαια και την Επιτροπή Γεωργίας για το γεγονός πως οι δικές μας προτάσεις ε, έγιναν αποδεκτές από το δικό σας προϋπολογισμό και νομίζω θα υπερψηφισθούν από την Ολομέλεια. Αυτό που με εκπλήσει είναι οι πρόσφατες αποφάσεις ε, του Συμβουλίου Γεωργίας γιατί αυτή τη στιγμή έξι κράτη-μέλη μπλοκάρουν την διατροφική, την επιστημιστική βοήθεια σε άτομα που την έχουν πραγματική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτής της ε, οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει ε, εκατομμύρια συμπολίτες μας δεν θα πρέπει να φανούμε άκαρδοι και θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Η κυρία Ράιμερς από την Επιτροπή Αλληλείας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, αξιότιμο Συμβούλιο. Στην Επιτροπή Αλληλείας ε, καταλήξαμε σε μια βιώσιμη ε, λύση, σε μια βιώσιμη διαπραγμάτευση που ε, φροντίζει στο να διατηρηθεί ο προπολογισμό όσο προβλέπετε. Είναι σημαντικό να έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα για να είναι η διαχείριση της αλίας βιώσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτελέσει τα καθήκοντά της και στο μέλλον σε ό,τι αφορά την πολιτική αλίας. Στέλνουμε μια δυναμική εξέλιξη. Και αυτό αφορά και τα πλητικά προγράμματα, την έρευνα, την διαχείριση των θαλασσών και σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι στην ε, ψηφοφορία να υποστηρίξετε τη γραμμή αυτή. Ελπίζω στις ε, διαπραγματεύσεις ε, τις επερχόμενες με το Συμβούλιο θα διατηρηθούν τα μέσα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ από την Επιτροπή Πολιτισμού ο κύριος Λόκιγκάρτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε σαν συντονιστή στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, με τα χαράς είδα ότι οι προτεραιότητές μας ελήφθησαν δεόντως υπόψη και θα ήθελα να ληφθούν υπόψη, δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη όμως. Την ίδια άποψη έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς, δηλαδή ότι χρειάζεται να επενδύσουμε σε τομείς που μπορούν να ευνοήσουν τα τηγική του 2020 και να δώσουν υπεραξία. Τα χρήματα που προβλέπονται για τη διαβίου ε, κατάρτιση είναι σημαντικοί ε, πόροι για την ανάπτυξη, πρέπει να διατηθούν και τα προγράμματα κινητικότητας όπως το Έρασμος και αυτό έχει στεφτεί με επιτυχία και πρέπει να υποστηριχθεί. Ο αθλητισμός έλαβε ένα ποσό που θα επιτρέψει να ε, υποστηριχθεί δεόντως και ελπίζουμε ότι τα αθλητικά προγράμματα θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν. Οι συνθήκες που καθορίστηκαν από την, Ευρωπαϊκή, από την Επιτροπή Πολιτισμού ε, καθόρισαν ότι πρέπει όσον αφορά την επικοινωνία να μπουν κάποιοι στο αποθεματικό. Η κυρία Κέλλερ για την Επιτροπή Ελευθεριών. Η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών χαίρεται που λαμβάνει περισσότερο για τη δικαιοσύνη και εσωτερικά και πολιτικέ ελευθερίε ένα μεγαλύτερο ποσό, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή η τομή είναι πάρα πολύ σημαντική για του πολίτε μα, για τι ελευθερίε του, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του σε συνολικό επίπεδο και να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Βεβαίω θέλουμε και εμεί να κάνουμε αυτό που πρέπει για να εξοικονομήσουμε χρήματα πιστεύουμε ότι πριν να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε καινούρια προγράμματα ή να παρατείνουμε να υπάρχοντα, χρειάζεται μια διεξοδική ανάλυση των υφισταμένων προγραμμάτων και θα πρέπει να μάθουμε από αυτά που συνέβησαν. Επιπλέον πιστεύουμε ότι οι δαπάνε θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη προστιθέμενη αξία πράγματι. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει νόημα να δημιουργούμε νέε υπηρεσίε ή να αναθέτουμε νέα καθήκοντα υφιστάμενε υπηρεσίε αν δεν έχουμε οικονομική βάση για κάτι τέτοιο. Μια υπηρεσία δεν μπορεί να πετύχει, να εκτελέσει καθήκοντα, άμα δεν έχει του αναγκαίου πόρου. Πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη όταν δημιουργούμε νέα προγράμματα και όταν καθορίζουμε, ε, δημιουργούμε μάλλον νέε υπηρεσίε. Ευχαριστώ, κυρία μου. Η κυρία Σιλβάνα Μέριν, Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Αναφορών το θέμα είναι η χρηματοδότηση του διαμεσολαβητή. Αυτό μας απασχολεί. Πρόκειται για ένα σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει αρρωγή στους Ευρωπαίους πολίτες και ε, προλαμβάνει σφάλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον προϋπολογισμό για το 2012 είναι πολύ συγκρατημένη η αύξηση για τον διαμεσολαβητή 0,4%. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις, δεν μπορούν να προσληφθούν νέοι υπάλληλοι. Το Συμβούλιο ήθελε ωστόσο να κάνει κάποιες περικοπές. Ευχαριστώ την Επιτροπή Προϋπολογισμού που δεν ενέκρινε τις περικοπές αυτές και ελπίζω σήμερα να επιβεβαιωθεί η θέση τη επιτροπή προπολογισμού. Αυτό θα αποτελέσει ένα μήνυμα για την εγκύτητα προ τον πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο και τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, οι ομιλητέ. Ο συνάδελφο, Λαβία από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι Υπουργέ, συνάδελφοι, Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τους συναδέλφους Μπαλζάνη και Φερνάντες ε, για την έξοχη δουλειά που έκαναν, την αξέπαινη δουλειά και όλους τους συναδέλφους για το πνεύμα συνεργασίας ε, που επεδείχθη φέτος. Έξοχη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις προτάσεις που έκανε στο σχεδίο προπολογισμού και η ερμηνεία που έδωσε το Κοινοβούλιο έδειξε ότι δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία των οριζοντίων περικοπών που ζητά το Συμβούλιο. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο ουσιαστικά μετέθεσε υποχρεώσεις και πληρωμές σε επίπεδο σχεδίου προπολογισμού. Να υπενθυμίσω ότι το επίπεδο 2012 είναι το έκτο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών. Δοθέντως αυτού θα πρέπει να εξετάσουμε εξ ολοκλήρου τις διάφορες στοιχές που αφορούν το επίπεδο των πληρωμών, δεδομένου ότι πολλά προγράμματα και δράσεις οδηγούνται προς το τέλος τους, εκπνέουν. Ε, θα πρέπει να δείξει την ε, υπευθυνότητα το Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, λαμβάνοντα υπόψη την κρίση που ζει η Ευρώπη. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξία μόνο για δύο κατηγορίε. μέσω επιλογής που βασίζεται επί τη δέουσα επιχειρηματολογία. Πάνω απ' όλα στην κατηγορία 4 ε, είδαμε ότι έγιναν διάφορα γεγονότα απρόβλεπτα στον αφορά την κατάσταση και χρειάζεται οικονομική υποστήριξη εκεί που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από το περιθώριο που έχει τεθεί τα θεματικά του 2012 και το 2α που ε, προτείνεται κατά 30,7 ε, εκατομμύρια ευρώ αύξηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού και χρηματοστικού συστήματος και να υποστηριχθούν οι πολιτικέ που έχουν προτεραιότητα το Κοινοβούλιο, που αντικαθρεφτίζουν και την στρατηγική του 2020. Πιστεύει ότι η ομάδα μα στιγμέ κρίσεω όπω είναι η παρούσα, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό θα πρέπει να είναι ένα μέσο επαναπροώθηση, να δημιουργεί πραγματικά προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκφράζω την ευχή το Συμβούλιο να μπορέσει να κατανοήσει την προσέγγιση που ακολουθήσουμε και να, να είναι ανοιχτό σε μια διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει συνεργασία και θα έχει σαν στόχο τον καθορισμό ενό προπολογισμού που θα είναι ρεαλιστικό και ο προπολογισμό που θα είναι για του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Γκόραν Φέρμ έχει το λόγο του SD. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφε, να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλσάνη, τον κύριο Φερνάντες και τον κύριο Ράιμερ Μπέγκε. Είναι πολύ καλή πρόταση Συχνά εμ, στην επικράτειά μου ακούω παράπονα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον φορολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι μόνο 2% των ευρωπαϊκών εξόδων προσρέουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ότι είναι μικρότερες οι αυξήσεις από τις εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει η εντύπωση ότι πάντα κάθε χρόνο γίνονται και επιστροφές στα κράτη-μέλη και δυστυχώς ότι πιστεύει ο κόσμος ότι χρειάζεται περικοπές ο ευρωπαϊκός προπολογισμό, αλλά ε, τότε θα είναι πραγματικά πιο δύσκολα τα πράγματα για τα πιο φτώχα κράτη-μέλη. Και ο Πολωνός ε, πρόεδρος υποστηρίζουν και άλλοι υποστηρίζουν την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Στην κατάσταση αυτή λοιπόν επιλέξαμε να είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες σε ό,τι αφορά την ε, προσέγγιση μας. Θέλουμε να γίνουν αυξήσεις μόνο σε τρει τομεί επενδύσει στην έρευνα, στην διαβίου μάθηση, διευθυντικά ταμεία στην Παλαιστίνη και στη Βόρεια Αφρική, προκειμένου να πετύχουμε μια προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουμε ε, την υπέρβαση της κρίσης. Πρόκειται για θετικές εξελίξεις. Χαίρομαι που συμφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ασφαλώς θέλουμε να υποστηρίξουμε και πολλά κράτη-μέλη. Θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση προκειμένου να μπορούμε να προασπίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε τους οικονομικούς τομείς. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κυρία Γένσεν. Sorry. Alde. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δύο εισηγητές, την κυρία Μπαλζάνη και τον κύριο Φερνάντες, για το πνεύμα συνεργασίας που δείξανε για τον προϋπολογισμό αυτό. Στην ομάδα μας θα δεχόμασταν να έχουμε κάποιες επιπλέον, ε, να έχουμε κάποια επιπλέον ε, πίπη αλλά για την κατάρτιση, για την έρευνα και για την εξωτερική πολιτική ε, νομίζω ότι εκεί θα είναι η τομή σου που θα πρέπει να εξετάσουμε, να δεχτούμε, με συγχωρείτε. Ε, ξέρω πως ε, κάποιες από τις περικοπές και προσπάθειες εξοικονόμησης που έκανε το Συμβούλιο είναι κάπως περίεργες, ε, κυρίως για την χρηματοδότηση κάποιων νέων οργανισμών κτλ. Μα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διανύουμε μια κρίση. πού θα κάνουμε λοιπόν τις οικονομίες ακριβώς στα μέσα τα οποία δημιουργούμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Νομίζω πως αυτό είναι αμφιβόλου επιτυχίας. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα και όχι ε, το θέμα των ε, πιστώσεων πληρωμών ε, ξεκομμένο από τις προτεραιότητες. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και ελπίζω πως ο διάλογος που θα γίνει θα είναι καθαρός ε, και βέβαια η Πολωνική Προεδρία έχει δείξει καλή θέληση. Καταλαβαίνω πως η θέση σας είναι δύσκολη. Ελπίζω όμως να βρούμε μια λύση η οποία θα επιτρέψει ο προπολογισμό μας να αντιμετωπίσει προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κύριος Μπόκρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση του ενδιαφέρον συζήτηση του προπολογισμού, ενδιαφέρονται οι αγορέ όσον αφορά την επιτόπιση τη κρίση του ε, ευρώ. Ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέλουν, πρέπει να ηγηθούν. Γενικά προσέχουν όλοι τι συζητήσει που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται ότι δεν έμαθε τα μαθήματα του περσινού έτου. Παρά τι τροπολογίε, εξακολουθούν να γίνονται απόπειρε για αύξηση των πληρωμών κατά 5% περίπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποφέρει και άλλη ήττα στο τέλο ε, Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερον, το να κάνουμε αύξηση του 4% του 5% όσον αφορά τις πυρομές και ανάληψη υποχρεώσεων είναι ένα χαστούκι προς τους πολίτες ε, ε, όταν τα κράτη-μέλη περνάνε ε, περίοδο κρίσης και εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας. Δείχνει έλλειψη σεβασμού έναντι των πολιτών και των χωρών που πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες. Και πρέπει να ζητούν οι φορολογούμενοι από τις Βρυξέλλες να κάνουν περικοπές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο για να σωθεί η Ευρωζώνη, αλλά όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και θα πρέπει να υποστηριχθούν επενδύσεις για το μέλλον. Όμως η υγιής διαχείριση του προπολογισμού θα απαιτούσε περικοπές σε άλλες κατηγορίες, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφείς αυξήσεις στις προτάσεις για τον προϋπολογισμό. Το δεν γίνονται αναγκαίε περικοπές από πλευρά Κοινοβουλίου. Προτείνει αυξήσει χωρίς να κάνει τις δέσου περικοπές αλλού. Το μοναδικό θετικό μήνυμα εν ώψη είναι η έκθεση Φερνάντες που σίγουρα προτείνει περικοπές σημαντικές στη μεταφράση και στη διερμηνία, στη διπορικά κλπ. Υποστηρίξαμε αυτέ τι τροπολογίε και ζητάμε και άλλε εξοικονομήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρίπελ για του πρασίνους. Κύριε Πρόεδρε Μπούζε, κύριε ε, Πίτρα Λεβαντόφσκι, κυρίε και κύριοι, ω ε, πολιτικό των Πρασίνων το βασικό κριτήριο για μένα είναι με του φυσικού πόρου να είμαστε προσεκτικοί και βιώσιμοι και ανάλογα θα πρέπει να διαμορφωθεί και προπολογισμό για να το πράξουμε αυτό και επίση ε, να είμαστε βιώσιμοι και σε ό,τι αφορά του χρηματοδοτικού πόρου. Αυτό μα το έμαθε η κρίση στην Ευρώπη. Και σε αυτό είμαστε σύμφωνοι και από τα τρία θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σχετική πολιτική. Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι επειδή όλοι είμαστε από κάποιο κράτο μέλο. Δεν είμαστε εξωγήινοι εδώ στι Βρυξέλλε. Καταλαβαίνουμε πόσο δυσχερή είναι η κατάσταση αλλά είμαστε πεπισμένοι ως ε, υπέρμαχοι της Ευρώπης ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την κοινή ευημερία των οικονομικών, στρατηγικών συμφερόντων μας και σε ό,τι αφορά την ευημερία των πολιτών μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ορθό ότι η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να τη λάβουμε πολύ στα σοβαρά και να επενδύσουμε πιο πολύ η βιωσιμότητα των νέων προϊόντων και νέων τεχνολογιών, η εξοικονόμηση σε θέματα ενέργειας, αποδοτικότητα σε θέματα ενέργειας, γιατί με τέτοια χρηματοδότηση των τομέων αυτών θα μπορέσουμε να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό επηρεάζει και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και γι' αυτό είναι σημαντικό από κοινού να προασπιστούμε αυτά τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό δεν είναι εχθρικό προς τα κράτη-μέλη, όχι, είναι στρατηγικά ευφυές να προασπιστούμε αυτή την ευρωπαϊκή υπεραξία προκειμένου να, να προωθήσουμε και την οικονομία των κρατών μέλων. Αφενός λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση αλλά και να επενδύσουμε ευφυώς σε κάποιους τομείς. Πού θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση σε επενδύσεις σε λάθος τομείς ε, για θέματα όπως για παράδειγμα στο ίτερ για την ατομική ενέργεια. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ξέρουμε πού πρέπει να προέλθουν και η πλειοψηφία του Συμβουλίου θέλει να χρηματοδοτήσει αυτή την επικίνδυνη τεχνολογία. Γιατί να μην κάνουμε εκεί εξοικονόμηση και πού άλλο να κάνουμε εξοικονόμηση στη διοικητική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην μετάφραση, στην διερμηνία 20 εκατομμύρια μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Θεωρώ ότι και στην πτήση business πρώτη θέση θα μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε σε πρώτη θέση. Ελπίζω να τα πετύχουμε αυτά. Ευχαριστώ και διακόπτει ο Πρόεδρο. Ο Μικέλ Πόρτα από την Ηνωμένη Αριστερά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο πρόβλημα με την πρόταση αυτή προπολογισμού είναι πως όσα έχουμε εντάξει εδώ αποφασίστηκαν το 2006. Δηλαδή μιλάμε για στοιχεία τα οποία προϋπάρχουν της κρίσης του 2008 και 2009, της κρίσης του χρέους. Άρα λοιπόν η πρόταση την οποία ε, συζητάμε δεν μπορεί ούτε να λύσει ούτε να αντιμετωπίσει την ε, κρίση την οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το 2012. Είναι πολύ περιορισμένος ο προϋπολογισμός για τις ευρωπαϊκές ανάγκες και οι κυβερνήσεις ε, μοιάζουν να έχουν πιστεί για το αντίθετο. Το δεύτερο πρόβλημα αυτής της πρότασης είναι πως υπάρχουν κάποιες ε, προϋπάρχουσες ε, ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για να εξυπηρετήσουμε κάποια μεγάλα συμφέροντα. Έχουμε ένα προϋπολογισμό που στηρίζει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτει την ασφάλεια και όχι την παιδεία ε, που δίνει περισσότερο στις φαρμακευτικές από ότι στην έρευνα ε, στα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να συγχαρούμε τους εισηγητές για τις προσπάθειες που κάνουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση αυτή προπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και δύο λόγια ε, για τα όσα έχουμε εντάξει εδώ στο κείμενο μας. Για πρώτη φορά κάνουμε μια προσπάθεια περιορισμού δαπανών και για το λόγο αυτό δεν κατανοώ γιατί έχουμε αφήσει εκτός αυτών των περιορισμών τις δαπάνες ε, των ε, ε, βουλευτών. Έχουμε μείωση 21% για διερμηνία και μετάφραση, κάτι το οποίο διακυβεύει θέσει εργασία, όπως επίσης δημιουργεί και προβλήματα για την πολυγλωσία. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό και δεν μειώνονται και τα γραμματι... οι, οι δαπάνες γραφείου για τους βουλευτές. Σε πολλά κράτη οι πολιτικές αυτές περιορισμού διερμηνίας και μετάφρασης έχουν ε, οδηγήσει σε μειώσεις μέχρι και 30% έχουν εγκαθεί θέσει εργασίας. Ε, είναι δυνατόν λοιπόν ε, εμείς απλώς να αφήνουμε τα δικά μας οικονομικά άθικτα και να προχωρούμε σε τέτοιου είδους οριζόντιες περικοπές. Τι θα πούνε οι συμπολίτε μας και πείτε μου πώς μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε τους συμπολίτε μας στα μάτια ε, κάνοντας κάτι τέτοιο. Ένα κοινοβούλιο το οποίο εξακολουθεί να, θεωρεί, να θεωρεί τα έσοδα των βουλευτών ε, να θεωρεί πως δεν μπορούν να θυγούν τα έσοδα αυτά των ε, βουλευτών. Καταλαβαίνετε πως η υπομονή των ε, συμπολιτών μας κάποια στιγμή θα εξαντληθεί. Η κυρία Μάρθα Αντρεάτσεν, πρόεδρε, πολλά κάτι μέλη πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα λιτότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε κατά 4,9% τον προπολογισμό του 2012. Αυτή η αύξηση δοθήσει της καταστάσεως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο, αλλά επέτρεψαν όμως αύξηση 2% που το θεωρώ απαράδεκτο. Το Κοινοβούλιο δεν άκουσε την πρόταση του Συμβουλίου και ζητά 5,2% αυξήσεις. Δικαιολόγηση για την αύξηση είναι η ανάγκη για επενδύσεις ούτως ώστε να βγει από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταματήστε. Σκεφτείτε. Διερωτηθείτε τι έγινε με τα χρήματα των φορολογωμένων που ήδη επενδύθηκαν για να επιτευχθεί ο στόχο ο μακρινό ε, του προγράμματο τη Λισαβόνα. Γιατί να διαθέσουμε σε αποτυχημένα προγράμματα χρήματα όπω το Γαλιλαίο που κοστίζει 22 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ στο φορολογούμενο ή προγράμματα όπω ο Ευρωπαϊκό Οίκο Ιστορία. Γιατί να μειώσουμε τι αμοιβέ των Ευρωβουλευτών. Και πάνω απ' όλα, πότε το Κοινοβούλιο θα σταματήσει να λέει αφήστε του να συνεχίσουν να ζουν όπω πριν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λούκα Χάρτονγκ για του μη εγγεγραμμένου. Πρόεδρε, έχω μια μεγάλη αίσθηση ντεζαβού σήμερα. Το Κοινοβούλιο και πάλι θέλει να αυξήσει τον προπολογισμό και πάλι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για εξοικονόμηση. Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει την κατάσταση, μάλλον καταφέρει να ζητήσει και πιο πολλά χρήματα από την Επιτροπή. Τρία εκατομμύρια για τους τουρκοκύπριους, ε, εκατομμύρια για τους εξωτερικούς οργανισμούς, 130 ε, ε, εκατομμύρια για project σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, 27 εκατομμύρια για αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Εμένη, Λατινική Αμερική και σαν κερασάκι στην τούρτα 100 εκατομμύρια για, επιπλέον για τις Παλαιστινιακές περιοχές. Είναι πραγματικά ντροπή του Κοινοβουλίου εδώ ε, να υπερψηφίσει αυτή την έκθεση. Θα έπρεπε να απαιτούμε πιο πολλά και αυτό καταδεικνύει μάλλον ότι δεν ε, λαμβάνουμε υπόψη τον πολίτη και το Συμβουλίο. Υπάρχει όμως ε, ένα φως στο τούνελ. Το αποτέλεσμα το σημερινό μάλλον η Ολλανδία μπορεί να εκφράσει το βέτο της. Ευχαριστώ άλλοι αγόριτες. Σαλβατόρ Γαρίγα Πολέδο, για δύο λεπτά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, την κυρία Μπαλσάνη, τον κύριο Φερνάντες, αλλά και τον κύριο Λαβία που μας παρουσίασαν με συνεκτικό και συνελετικό τρόπο θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και έχουν ε, προκαλέσει συγκρούσεις μέσα στις πολιτικές ομάδες. Τώρα, ε, για να εκφράσω τα όσα πιστεύει η δική μας ομάδα, εδώ πέρα έχουμε συνδυάσει την απαραίτητη λιτότητα με την επαρκή χρηματοδότηση και για την ανάληψη υποχρεώσεων και για τις πιστώσεις πληρωμών. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις ροφές των διάφορων ε, θέσεων και νομίζω σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει και εξασφαλίζουμε και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο όπως επίσης και την πολιτική γειτονία. Άρα λοιπόν πιστεύω πως εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Τώρα για το ίτερ η χρηματοδότηση είναι πρόβλημα του μέλλοντος, είναι πρόβλημα της τρέχουσας περίοδου. Η ομάδα μας δεν μπορεί να δεχτεί πως ο προπολογισμό ε, του 2012 θα αλλάξει πάρα πολύ λόγω της θέσης του Συμβουλίου εδώ. Τώρα για τις πληρωμές ε, περιμένουμε τι θα γίνει στη συνδιαλλαγή. Αλλά θα πρέπει το Συμβούλιο και εδώ να δει τι θα γίνει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει έναν διορθωτικό προϋπολογισμό ο οποίος θα κατατεθεί στα τέλη της χρονιάς. Αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ε, πιστώσεων από αυτή που αναμένεται. Ίσως λοιπόν το να αφήσουμε στο 2% ε, όπως προτείνει το Συμβούλιο δεν θα σε επιτρέψει να διατηρηθεί η πολιτική έρευνα ή συνοχής για το 2012. Νομίζω λοιπόν πως για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζει έναν πραγματικά ε, σφιχτό προϋπολογισμό και έχουμε θυσιάσει αρκετά. Ε, για παράδειγμα, έχουμε, μειώ, έχουμε παγώσει ε, τα οδηπορικά, έχουμε μειώσει τα οδηπορικά και τις, τα διάφορα επιδόματα στους βουλευτές. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαρίδο. Τώρα έχει το λόγο για, μισό, για 1,5 λεπτό ο κύριος Βόν. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εισηγητές και καλωσορίζω την προσέγγιση που ακολουθήθηκε που μείωσε την αύξηση στο 0,8%. Καλωσορίζω ιδιαίτερα το πάγωμα των, ε, των γενικών εξόδων 2012, 5% περικοπές όσον αφορά τα οδηπορικά εξοικονομήσεις στο κόστος μετάφραση και διερμηνία και όλες άλλε άλλες οικονομίες που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων. Βεβαίω η ομάδα S&D ίσως θα ήθελε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και γι' αυτό υποβάλαμε τροπολογίες που ζητούν ένα πάγωμα σε όλε τι αποζημιώσει και τι ημερήσιες αποζημιώσει για το 2012. Ζητήσαμε το Προεδρείο να ε, κάνει με εξολόγηση των διπορικών και να βρει τρόπους για την μείωση του αριθμού των ε, εισιτηρίων business και ζητούμε να γίνει συγκριτική μελέτη του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκρίνοντα το δικό μα προπολογισμό με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ζητήσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική για τα κτίρια και ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται στο μέλλον Πλήρω για προτάσεις για νέα ε, κτίρια. Και προσωπικά θα ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο από αυτό και να ζητήσω για ένα πάγωμα σε όλες τις ε, αποζημιώσει και αμοιβέ για το υπόλοιπο αυτή τη θητεία, διότι είμαι σίγουρο ότι με περισσότερη δουλειά, με περαιτέρω ανάλυση των δαπανών του Κοινοβουλίου, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και να κάνουμε ακόμα περισσότερε οικονομίε. Κάναμε καλή αρχή φέτο ε, δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομίες και ταυτόχρονα μπορούμε να προστατεύσουμε και τη σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Άλβαρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε, καλημέρα και προς την Προεδρία του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι ο εισηγητής Φερνάντες ε, σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό το προπολογισμό του προπολογισμού πέτυχε κάτι πολύ καινούριο, αν θέλετε, μια καινοτομία για τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι που ήταν στενή συνεργασία. Σε καιρούς που πρέπει να σφίξουμε τις ζώνες και εμείς ε, συμβάλαμε ότι μπορούσαμε για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων. Νομίζω ότι αποτελεί αυτό ένα σημαντικό μήνυμα σε καιρούς που όλα τα κράτη-μέλη συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν την κρίση. Νομίζω ότι δώσαμε το καλό παράδειγμα. Κάναμε εξοικονόμηση 47 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συνάδελφος Βόν μας ανέφερε τα σχετικά ποσοστά, αλλά σίγουρα ε, μπορούμε να κάνουμε και περαιτέρω εξοικονόμηση. Δεν πρέπει απαραίτητα να αγοράσουμε κτίρια 30 εκατομμυρίων ευρώ θεωρώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους μας και επίσης θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη οικονομία για την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική διαχείριση. Αν η Επιτροπή Προϋπολογισμού δεν ε, ε, λαμβάνει μόνο τις γραμμές που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά έχει μια γενική επισκόπηση για να μπορεί να δει πώς δαπανώνται τα σχετικά μέσα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πενταπλάσιες οικονομίες αν δεν πηγαίναμε, ερχόμασταν κάθε μήνα στο Στρασβούργο, αλλά μέναμε στις Βρυξέλλες για την Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άλμαρο. You just in time. Φτάσατε την κατάλληλη στιγμή, κύριε Έλλης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω τα όσα στηρίξει η ομάδα μου σήμερα το πρωί. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε και κάποιες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του 2012 γιατί πολύ σωστά στη συζήτηση μέχρι σήμερα εστιάσαμε στο ποιες είναι οι προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως στο συγκεκριμένο πλαίσιο που ζούμε με τις μεγάλες ε, συζητήσεις που γίνονται στην Ήπειρό μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους, πως ε, στη συγκεκριμένη διαδικασία για το 2012 δεν έχουμε εστιάσει ιδιαίτερα το βλέμμα μα στο πού θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια στον προπολογισμό έτσι ώστε να βρούμε και κάποια να απελευθερώσουν κάποια κονδύλια για προτεραιότητες που θα έχουν στο μέλλον θεσπιστεί, για παράδειγμα έρευνα κτλ. Στη διαδικασία λοιπόν του προϋπολογισμού θα έπρεπε να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομία μέχρι 2 δις ευρώ. Όπου γραμμές, για παράδειγμα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Εκεί πολλές φορές μπαίνουμε σε συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο και πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πού δαπανούμε ε, κονδύλια με τρόπο ο οποίος δεν είναι αποτελεσματικός. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Αλφόνση έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ομάδα μας τα απόσχει από την ψηφοφορία. Αυτή η αποχή είναι αποτέλεσμα αντιφατικών συναισθημάτων. Από τη μία πλευρά δεν μπορούμε να καταγγείλουμε την αδράνεια ε, και όσον αφορά τα ενεργειακά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την προηγούμενη συζήτηση του προπολογισμού είχαμε την πυρηνική καταστροφή τη Φουκουσίμα. Η Γερμανία, η Ιταλία, ε, η Ελβετία και άλλοι ε, έμαθαν τα βασικά μηνύματα. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εκφράζει ο προπολογισμό, τίποτα δεν κινείται, σχεδόν τίποτα. Κάποιε μικροπροσαρμογέ όσον αφορά το αποθεματικό και πάντα αυτή η αιμονή υποστήριξη οικολογικών και τεχνολογικών αδιεξόδων, όπω το αέριο από το σχιστόλιθο και το πρόγραμμα η ΤΕΡ που κοστίζει πολύ και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πλειοψηφία για να αντισταχθούμε στις μεγάλες περικοπές που ζητά το Συμβούλιο. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις πληρωμές ενώ ε, λύγει το έτος του 2012 και προς το τέλος του 2007-2013. Και ε, δεν είναι ένα μέτρο οικονομίας που μας προτείνει το Συμβούλιο, είναι ένα μέτρο στραγγαλισμού το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αλληλέγγυο έναντι αυτή αντιευρωπαϊκή ε, στάσεω. Τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει, είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι ο προπολογισμό ευρωπαϊκό ποτέ δεν ήταν ελληματικό, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό χρέο και ότι δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία μέσω του κοινή χρήση των πολιτικών και των μέσων. Η επίθεση κατά των οικονομικών μέσων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι η καταπολέμηση οικονομική μοτοστική κρίση, θα είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κλούτε. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μένει λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Αλλά επειδή διαφρύνονται οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργήθηκαν στις δημοσιονομικές προοπτικές νέες υπηρεσίες. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται σωστή χρηματοδότηση μετά την χρηματοπιστωτική τραπεζική κρίση αναδείχθηκαν οι αδυναμίες κάποιων κρατών μελών και μάλιστα με κατεπίγοντα τρόπο για την ενίσχυση των κρατών αυτών θα χρειαζόταν ένα οικονομικό πρόγραμμα. Κάποιοι ειδικοί μιλούν για την αναγκαιότητα ενός σχεδίου Marshall για την αντιμετώπιση της κρίσης σε κάποιες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ε, ανάπτυξης για τους επιχειρηματίες, για τους ε, νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τι έρχεται και κάνει το Συμβούλιο, κάνει περικοπές στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα πολιτική κατάσταση, η αύξηση του, του προπολογισμού, αν θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί αύξηση του προπολογισμού, τουλάχιστον θα πρέπει να προασπιστούμε τον υπολογισμό και να μην αφήσουμε να γίνουν περικοπές που προτείνει. Ευχαριστούμε κύριε Κλούτη. Ο κύριος Μοργάντη έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι μια στιγμή οικονομική κρίση και τώρα θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένε απαντήσει η Ευρώπη και είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία πέρα από την αύξηση του προπολογισμού που φαίνεται κάτι υπερβολικό. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν περικοπέ από τι σπόρο γενικομισέ επιχειρήσει από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό το αποτέλεσμα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Το Frontex είναι άλλη σημαντική πτυχή. Το Συμβούλιο έκανε λάθο ε, να, δώσει νέε εξουσίε χωρί επαρκή Επ' αυτού και από όλου του θέματος που αφορά τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι είναι πολύ πιο υπεύθυνο. Αυτό είναι σίγουρο. Όσον αφορά τις περικοπές, παραθέσει τα διπορικά ε, του Κοινοβουλίου ε, ε, η πραγματική οικονομία θα ήταν να εξαλείψουμε το Στασβούργο. Οι συνθήκες θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και αυτές οι δύσκολες συνθήκες τελικά θα έπρεπε να επαναξεταστούν και να εξεταστεί και το θέμα της έδρας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοργάντη. Θα δώσω τώρα το λόγο για ένα λεπτό στην κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η βασική γραμμή του ΕΛΚ σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2012 είναι τα μέτρα να εστιαστούν στην επίτευξη της στρατηγικής ε, για το 2020. Ο προπολογισμό για το 2012 ε, έχει μειωθεί γιατί έχουμε πιο πολλά έξοδα για τα 18 νέα μέλη τα οποία υπολογίζονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και σε ό,τι αφορά την προσχώρηση της Κροατίας. 1,9% σε σχέση με το 2011. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για την πιο χαμηλή αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια. Ήδη τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να προσθέσουμε νέες, νέα καθήκοντα και νέες αρμοδιότητες χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, όπως για παράδειγμα την προσθήκη των, νέων, των τριών νέων ε, υπηρεσιών για τις χρηματοπιστωτικές, χρηματοπιστωτικές αγορές. Θεωρώ ότι αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η ενιαία αγορά και η επένδυση στην ε, εκπαίδευση της νεολαίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις συναδέλφους, τους τρεις εισηγητές των εκθέσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμασούρ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ του εισηγητέ για την εξαιρετική του δουλειά και να πω κάτι συμπληρωματικό. Πριν από δύο χρόνια πριν από μόλι δύο χρόνια και κάποιοι συνάδελφοι δείχνουν ότι έχουν ξεχάσει, οι Υπουργοί Οικονομικών κατηγορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, χρηματοδοτεί λίγο και αργά. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον ε, ε, ηρωνικό το ότι προσπαθεί τώρα το Συμβούλιο να μπαλώσει τις τρύπες προπολογισμού και στο χρέος που δημιούργησε αυτή η προσέγγιση. Είμαστε αυτή τη στιγμή και αναγνωρίζουμε απόλυτα ε, τους περιορισμούς στους οποίους δεν μπορούν να αποφύγουν πλέον οι εθνικοί προϋπολογισμοί και αυτό φαίνεται από τις πιστώσεις πληρωμών. Θέλουμε να φτάσουμε σε μια γρήγορη ε, συμφωνία. Αλλά υπάρχουν διάφορα σημεία. Καταρχήν, πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Το είπαν οι συγγητέ. Και κυρίω τι γίνεται ε, με, ε, με τι πληρωμέ για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και για να ενισχύσουμε τη θέση τη Ευρώπη. Δεύτερον, συνέπεια μεταξύ των αποφάσεων του Συμβουλίου και του τρόπου που τοποθετούνται ω πιστώσει στον προπολογισμό. Για παράδειγμα, μεταναστευτική πολιτική ή χρηματοπιστωτική εποπτεία θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε την δικαιοσύνη για τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την ευρωπαϊκή βοήθεια για να καλύψουν την ε, καθυστέρηση στις οποίες τις καταδίκασε μια άδικη ιστορία. Είναι τα έμεσα θύματα της κακοδιαχείρισης άλλων κρατών μελών. Και τέσσερα, η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων των δράσεων που έχουμε στην Ευρώπη 2020 για το ΦΑΡ. Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή κατανοούν πως ο μόνος τρόπος να καλύψουμε το χρέος μας είναι να γυρίσουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Δεν θα πρέπει να τυφλωθούμε όταν ε, ε, βλέπουμε πως οι άλλοι έχουν αρχίσει να βρίσκουν το φως τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασούρ. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Χέρτζοκ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μπαζάνη και τον κύριο Μανουέλ Φερνάντες ε, και τον κύριο Μπέγκερ να πω πρώτα απ' όλα κάποιε παρατηρήσει. Να, μην χρειαζο... να μην έχουμε περισσότερα χρήματα, χρειαζόμαστε όμω ισχυρότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ισχυρότερη ενιαία αγορά, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη περιφερειακή ενίσχυση, περισσότερη ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι δαπάνη, αλλά επένδυση. Επένδυση για το μέλλον επένδυση για τις οικονομίες των κρατών μελών. Και έτσι μπορούμε να πετύχουμε ευφυή, βιώσιμη, ενταξιακή ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η πραγματική μάχη κατά της φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιμείνει από αυτού κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής δεν πρόκειται να αρχίσουμε παζαρέματα που θα υπονόμευαν του στόχου Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Κοινού στόχου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χάκλουν, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εισηγητές, οι οποίοι έκαναν πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Προσπαθήσαμε στις διαπραγματεύσεις που ήταν πάρα πολύ δύσκολες να σημειώσουμε πρόοδο. Αλλά το επίπεδο δαπανών που έχουμε πλέον μπροστά μας είναι κάτι το οποίο δεν αποδέχονται τα κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει ότι από κοινού θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό, σε μια κοινή θέση για το 2012. Ήμουν υπεύθυνο εξ ονόματο των φιλελευθέρων και προτείναμε για παράδειγμα να γίνουν περικοπές. Δυστυχώς, στην ψηφοφορία δεν επικράτησαν αυτέ οι απόψει. Και γι' αυτό λοιπόν θα απόσχουμε σήμερα. Θετικά όμως έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Θέλουμε για την Ευρώπη του 2020 να επενδύσουμε σε ό,τι αφορά την στρατηγική αυτή. Ε, δαπάνε στην έρευνα, στην κοινοτομία, στην παιδεία. Α, παράλληλα διαπιστώνουμε ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει την ε, απεριόριστη αύξηση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού θα κάνουμε καινούριε δαπάνες, αλλά και πού θα κάνουμε οικονομίες. Εμείς θα θέλαμε η συζήτηση να ήταν πιο επικοδομητική σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες περικοπές. Δεν τα καταφέραμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Έπινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ζητούμε από τους, τους ε, πολίτες να σπίξουν τις ζώνες. Και αυτοί μας ρωτάνε τι κάνετε εσείς. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, αλλά δεν κάνουμε καθόλου ε, δεν ασκούμε καθόλου πολιτική λιτότητα. Αντιθέτως, αυξάνουμε τον προπολογισμό. Μέχρι πρόσφατα, οι περικοπές στον προπολογισμό θεωρούντουσαν αντιευρωπαϊκέ, αλλά στι παρούσε συνθήκε είναι μάλλον υπέρ τη Ευρώπη ε, ω τακτική. Ω μέλο του ECR, πάντα πρότεινα να αναθεωρηθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον κύριο Φαν Όρντεν καταρτήσαμε μια μελέτη σε ό,τι αφορά την περικοπή ε, κατά 25% του προπολογισμού. Έχω αποστείλει αυτή τη ε, μελέτη που ονομάζεται Ending the Access ε, στα μέλη των επιτροπών. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το γλωσσικό καθεστώς, να περιορίσουμε τον αριθμό των γλωσσών σε ό,τι αφορά τη μετάφραση στα προπαρασκευαστικά στάδια και θα πρέπει να κοιτάξουμε προγράμματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ και ε, κάνουν τους πολίτες να μας μισούν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Έπιν και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Φανέκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα που όλη η Ευρώπη πλήγεται από μια σοβαρή κρίση, καταρτίζουμε έναν εξευτελιστικό προϋπολογισμό. Εξευτελιστικό γιατί δεν κάνουμε καμία σοβαρή προσπάθεια να κάνουμε σοβαρή οικονομία καταργώντας κάποιες τελείως άχρηστες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και έχω υπόψη μου για παράδειγμα την Επιτροπή Περιφερειών, την ΕΟΚΕ, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι χρησιμότητα εξυπηρετούν και όλα αυτά κοστίζουν 250 εκατομμύρια στον φορολογούμενο κάθε χρόνο και να μην αναφέρω τα 9 εκατομμύρια το χρόνο για την ε, ευρωπαϊκή τηλεόραση, 3 εκατομμύρια που χαρίζουμε στους ε, Τούρκους ε, που κατέχουν την Κύπρο και άλλες τέτοιες εξευτελιστικές πρακτικές. Δεν καταφέρνουμε ούτε και το ίδιο με τις αποζημιώσεις, τις αμοιβές να τις κρατούμε σε λογικά επίπεδα και με αυτή την υποκριτική πολιτική θα πρέπει να σταματήσει για να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες μας ότι ακόμα και εμείς οι προνομιούχοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Συζητάμε αυτή τη στιγμή τον προπολογισμό του 2012 και σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ε, Βρυξέλλες συζητά τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Είναι περίεργο κάπως να ψηφίζουμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό στήριξης. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα. Έχουμε κρίση, λείπουν θέσεις απασχόλησης, μιλάμε για ανάγκη επενδύσεων. Ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός πρέπει να είναι επενδυτικός προϋπολογισμός, στο 95% τουλάχιστον των όσων προτείνει. Χρειάζονται ευρωπαϊκές υποδομές στην ενέργεια, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές. Θα πρέπει να επενδύσουμε και εδώ. Είμαστε η πιο στεναρή παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει επιτέλους να κλείσουμε όλα τα θέματα στην ενιαία αγορά και θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να παίξει το ρόλο του ε, γιατί έχουμε θεσπίσει προτεραιότητες στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Η παιδεία, η έρευνα, θα πρέπει μέσω του προπολογισμού να τους κατακτήσουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία προσφέρουν περισσότερο και υπάρχουν άλλα που έχουν μικρότερη συμμετοχή. Ε, δεν έχουμε όλη την ίδια κλίδα κατανομής ε, για να ακολουθήσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά, ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις του προπολογισμού. Δηλαδή για κάθε ευρώ που επενδύεται σε ένα κράτος μέλος, ποιο, τι τι προσφέρει στο κράτος μέλος αυτό, ποιο τμήμα ενός ευρώ, ενός ευρώ παραμένει στο κράτος μέλος. Ε, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προετοιμάσει μια τέτοια μελέτη. Πιστεύω πως το ευρώ που επενδύουμε σε μια νέα περιοχή, σε μια ευρωπαϊκή περιοχή, επηρεάζει και όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός προετοιμάζει το μέλλον μας και θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Το μέλλον μας εξαρτάται από το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας αφήσουμε στην άκρη τους λαϊκισμούς και ας ψηφίσουμε τον προπολογισμό όπως έχει μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γκαλτιέρη για ένα λεπτό. Το κεφάλαιο 4 υποχρηματοδοτείται συστηματικά εναντί των δεσμεύσεων και στοτικών στόχων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και αυτό μα οδήγησε σε πόδινε επιλογέ για να διαφυλάξουμε τι προτεραιότητέ μα και πιο συγκεκριμένα του πόρου για την Παλαιστίνη, που προφανώ είναι αναγκαίοι πόροι, κυρίω υπό το φω των επιλογών του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ οι περικοπές μετά στην ΚΕΠΑ που δεν είναι μάλλον γενικές περικοπές αλλά πολιτικές περικοπές σε συγκεκριμένο σημεία που δεν επηρεάζουν τις άλλες επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα το Αφγανιστάν περικοπή επώδυνη αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι παρά τα καλά αποτελέσματα των αποστολών μας σε, αυτή σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμπροματικός φορέας που υπόκειται στρατηγική άλλων και πληρώνει περισσότερο. Δεν υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Κατεπήγονται μέτρα το πρόβλημα των ειδικών απεσταλμένων. Εδώ είναι μια περικοπή που έχει μια λογική. Προπαρασκευαστικά μέτρα το Συμβούλιο αρνείται το άρθρο 51 ε, του Δημοσιονομικού Οργανισμού που δίνει περιορισμένο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τη τη Συμφωνία τη Μαδρίτη. Άρα εδώ είναι οι περικοπέ αναπόφευκτε. Δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επέλεξε αυτή την γραμμή τη λιτότητα. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να εκφράζει λοιπόν απορίες όσον αφορά τι συνέπειε αυτή. Δεν είναι η κυρία Ζεντρεζεύσκα στην αίθουσα, άρα λοιπόν θα δώσω στην κυρία Γκρελιέ το λόγο για ένα λεπτό. Για δεύτερη χρονιά βλέπουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση προπολογισμού επιτρέπει με τα βία να εφαρμοστούν τα προγραμματισμένα προγράμματα χωρί να λάβουν υπόψη τι αρμοδιότητε τη Λισαβόνα. Στο δόγμα τη λιτότητα βασίστηκε το Συμβούλιο και αποφασίζει αυθαίρετε περικόπε όσον φορά τα προγράμματα που έχουν στη σημασία εν ώψη του οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου. Ε, Εμεί θέλουμε να κινητοποιήσουμε το, ε, στη στρατηγική του 2020 του προπολογισμό και τονίζουμε τα προγράμματα που αφορούν την έρευνα, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, την συνοχή, τι επενδύσει, τι δημόσιες. Είναι μια θέση συνεπή που θα πρέπει ε, να αναγνωρίσουμε ότι υποστήριξε η κυρία Μπαλζάνη στην έκθεσή τη. Ο ε, προπολογισμό ε, δεν πρικοδοτείται παρκώς. Τα κράτη-μέλη έχουν μόνο τη λιτότητα σαν στόχο. ο δημόσιο τομέα περιορίζεται. υπάρχει μακροοικονομική ρεσιμότητα που επιβαρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση και πλήττονται οι πιο ευάλωτοι πολίτε. Και έχει επιφυλάξει και τη συνεπιστική βοήθεια κακή μοίρα το Συμβούλιο. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν οι ίδιοι πόροι επαρκή, δεν υπάρχουν ευρωομόλογα, μια δικυβερνητική μέθοδο κυριαρχεί και ένα προπολογισμό είναι γελίο. Όπω και αυτή η συζήτηση εν ώψη των διακυβευμένων τη Συνόδου Κορυφή τη Ευρώπη και ε, ο Σαρκόζη και η κυρία Μέρκελ προσπαθούν να διαθέσουν δισεκατομμύρια για να σώσουν τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανλίστερ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να περιοριστώ σήμερα σε ένα τμήμα τη χρήση του μέσου ευελιξίας για το 2012 για δύο σκοπούς την ε, πολιτική γειτονία και την έρευνα και την ανάπτυξη. Και τα δύο αυτά σημεία έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι μάλλον και διαπιστώνουμε μεγάλες ελλείψεις στην ε, εκτέλεση την ε, Κυριακή έγιναν οι εκλογές στην την Ισία ε, και το είδα από κοντά γιατί ήμουν μέλος της αποστολής. Ε, χρειάζεται η αραβική ανάπτυξη συγκεκριμένη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον συνεχή εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη και το 7ο πρόγραμμα ανάπτυξης. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρόκειται για κάτι βασικό για την οικονομική ανάκαμψη. Το μέσο ευελιξίας Μα δίνει τη δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα προς υποστήριξη αυτών των δύο προτεραιοτήτων και εξ του ΕΛΚ. Απευθύνουμε έκκληση προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσει προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Φανίστηλ Ρόι και τώρα ένα λεπτό. Η κυρία Καρία Θάμπα Λουρβιάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Ζούμε σε συνθήκες κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό πρέπει να βρούμε ένα εργαλείο στήριξη όλων των κρατών. Θα πρέπει να θεωρήσουμε πως είναι ένα μέσο που εξασφαλίζει αλλά και αυξάνει τις πολιτικές σε δημόσιες επενδύσεις. Γιατί με τον προπολογισμό αυτό διατηρούμαστε στο επίπεδο ε, χρηματοδότησης βασικών ε, πολιτικών όπως η κοινή γεωργική, η κοινή εργοδοτική πολιτική, ε, η πολιτική συνοχής. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους παραγωγούς, στους οποίους έδειξε η κρίση ε, με τα e. για παράδειγμα. Ε, μέσα στον προπολογισμό αυτό βλέπω πως τονίζουμε την ανάγκη που υπάρχει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ακολουθήσουμε μια πολιτική βιώσιμης και αλληλέγγυας ανάπτυξης και εφιούς ανάπτυξης το Εράσμο λοιπόν η διαβίου μάθηση, η νεολαία σε κίνηση ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθούν από την πρότασή μας και βλέπω πως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την Παλαιστίνη και την πολιτική γειτονία γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αραβική άνοιξη. Ζητώ λοιπόν από το Συμβούλιο να κάνει μία ακόμα προσπάθεια και να στρατευθεί έτσι ώστε να έχουμε μία Ευρώπη πιο φιλόδοξη στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκάρτια Σάβαλ. Φαίνεται πως η κυρία Γεντρεζεύσκα έφτασε. Θα σας δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω πως ακριβώς όπως πέρσι, έτσι πάλι και φέτος, ε, περιμένουμε να κάνουμε κάποιες δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό του 2012. Νομίζω πως εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ποιες είναι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι ζωτική σημασίας και εξασφαλίζουν τη συνέχεια σε σχέση με τα όσα έχουμε κάνει περασμένα χρόνια. Δηλαδή, θα ήθελα να ε, υποστηρίξω το πρόγραμμα διαβίου μάθησης της νεολαίας σε κίνηση Youth in Action, όπως επίσης και, και ολόκληρο ε, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση στο Συμβούλιο. Θα ήθελα τις τροπολογίες τις σχετικές να τις κρίνετε θετικά και με κατανόηση να δεχτείτε τις προθέσεις αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ως σκοπό να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην καινοτομία, ε, στις ευκαιρίες για τους νέους, ε, δεδομένης και της ανεργίας ε, των νέων, μια και ξέρουμε όλοι πως είναι πολύ δύσκολο για τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι ευρωπαϊκές πολιτικές ποτέ δεν θα είναι επαρκής. Αν όμως υπερψηφίσουμε αυτή την αύξηση, νομίζω ότι με σαφήνεια θα υποδείξουμε ε, το δρόμο τον οποίο θα θέλαμε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ε, της απασχόλησης ε, και της ανάπτυξης. Νομίζω πως η θέση μας για την αύξηση της πολιτική συνοχής θα πρέπει να στηριχθεί. Το ξέρω πως το κάνει το Κοινοβούλιο, θα το κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να το κάνει και το Συμβούλιο, γιατί εκεί θα έχουμε πολλέ πληρωμέ του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεντριζεύσκα. Νομίζω ότι φτάσαμε ε, στο Catch the Eye. Θα δώσω πρώτα απ' όλα τον κύριο, στον κύριο Αμπάτ το λόγο με τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σε ένα πλαίσιο οξία κρίσεω και έχουμε ισορροπημένο προπολογισμό και υπεύθυνο που καθορίζει κάποιε προτεραιότητε. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα, αμοιβαιότητα όσον αφορά τι διεθνεί συναλλαγέ ε, των παραγωγών, αλλά χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική και πολιτική ενέργεια και έρευνα που θα είναι ισχυρέ και χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να μιλά με μια φωνή στον κόσμο. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίση ένα προπολογισμό, όπω υπενθύμησαν και κάποιοι συναδέλφου μου, ένα προπολογισμό που διατηρεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα άτομα που έχουν ανάγκη και το πρόγραμμα τη Ευρώπη για την νεολαία, που είναι η πρώτη στην κρίση, αυξάνοντα κατά 5% την υποστήριξη για τα προγράμματα lifelong ε, learning, δίνουμε ένα σημαντικό μήνυμα Δηλαδή ότι θέτουμε την κινητικότητα, τη θελοντική συμμετοχή και την αλληλεγγύη σαν φορεί αλλαγή για του νέου στην Ευρώπη. Με το πρόγραμμα η, νεολαία σε και μπορούμε να εμβαθύνουμε δημιουργώντα ένα πραγματικό έρασμο τη μαθητεία. Όσον αφορά την κρίση, χρειαζόμαστε πραγματικό ομοσπονδιακό προπολογισμό με ιδίου πόρου, όπω η φορολόγηση των συναλλαγών, κάτι που πρότεινε ο πρόεδρο Σαρκοζή και η καγκελάριο κυρία Μέρκελ. Σε διεθνέ κλίμα που γίνεται όλο και πιο δύσκολο, θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και να κάνουμε εργαλείο προπολογισμό που θα βοηθήσει την Ευρώπη και του πολίτε και να ενοποιήσει τελικά και να προωθήσει την Ευρώπη των παραγών. Ευχαριστώ κύριε Μπάτ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπαλσίτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ περίπλοκη σήμερα και οι προσπάθειές μας να πετύχουμε συνένεση όταν συζητούμε τον προϋπολογισμό του 2012 χρειάζεται τεράστιες προσπάθειες. Ευχαριστώ τη συνάδελφό μου, την κυρία Φραντσέσκα Μπαλζάνη και τους άλλους που συμμετείχαν στην σύνταξη της πρότασης. Προσβλέπουμε σε μια απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί στις Βρυξέλλες, όμως όποια, πρόταση, απόφαση και αν ληφθεί θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Συνεπώς ο προπολογισμό του 2012 μπορεί να είναι ιστορικό προπολογισμό. σω επιτρέψει στην Ευρώπη να σταθεροποιηθεί. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, όπω ανέφερα και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να μην μειώσουμε τι επενδύσει στην καινοτομία και την έρευνα θα πρέπει να επεξετάσουμε την αγροτική πολιτική, του ώστε στο μέλλον όλα τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούνται ισοδίκαια σε αυτό το τομέα, να εξασφαλίσουμε και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Πρωταρχικό στόχο βεβαίω είναι αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Εκεί θα πρέπει να συστηθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές, την κυρία Μπαλτσάνη και τον κύριο Φερνάντες και τον Σκιώδη τον κύριο Λαβία για την έξοχη δουλειά που έκαναν επί ενός προπολογισμού για το 2012 που αντιπροσωπεύει μια επιτυχία για αυτό το κοινοβούλιο παρά τις δυσκολίες για την επίτευξη ε, του ελάχιστου επίπεδου αυξήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λιτότητας που επικρατούν αυτή την περίοδο για πρώτη φορά ο προπολογισμό του 2012 επικεντρώθηκε επί των στόχων των συγκεκριμένων και προτεραιότητε όσον αφορά του νέου, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την έρευνα και την καινοτομία. Είναι Αν εισηγήτρια του προπολογισμού τη Επιτροπή Γυναικών, πρέπει να πω ότι έχω ικανοποιηθεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Δάφνη που υποστηρίζει τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ήταν κάτι που ε, επανήλθε στα επίπεδα πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων ε, κράτησε τα επίπεδα χρηματοδοτήσεων που βλέπει το σχέδιο προπολογισμού. Οπότε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους ηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματέρα. Ο κύριος Φαν Ντάλεν έχει το λόγο. Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το αύξηση του προπολογισμού δεν πρόκειται να την στηρίξω. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θέλει να αυξήσει κατά 4% τις δεσμεύσεις και 5% τις πληρωμές. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε όπου ε, καταρτίζονται προγράμματα λιτότητας ε, και να εξισορροπηθούν οι προϋπολογισμοί το Κοινοβούλιο κλείνει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα και συνεχίζει στην τάση των προηγούμενων ετών, αυξάνοντας διαρκώς τον προπολογισμό. Σε ένα τμήμα, θεωρώ ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, η Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, υιοθέτησε μια πρότασή μου για την, ε, το πάγωμα 15% των ταξιδιωτικών εξόδων. Θα πρέπει να, δείξει, να καταδείξει ο Γενικός Γραμματέας πρώτα ότι χρειάζονται πραγματικά πιο πολλοί πόροι. Και την άνοιξη θα αποφασίσουμε κατά πόσον θα διαθέσουμε ή όχι το 15%. Θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να καταστεί ε, πρακτική συνηθισμένη σε κάθε διαπραγματεύση του προπολογισμού, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο προπολογισμό που έχουμε μπροστά μας για μια φορά ακόμα αποδεικνύει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. 0,8% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολυετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε ε, θεσπίσει ε, και προσπαθούμε με τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας να εξασφαλίσουμε κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ξέρετε πως αυτή τη στιγμή τρέχουν ε, προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και ζούμε στην Ευρώπη της διαφοράς, όχι της ομοιότητας και αυτό φαίνεται από τον προπολογισμό. Εάν εμείς θέλουμε να σεβαστούμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε ένα ε, προπολογισμό που θα επιτρέψει την επανακεφαλοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ε, θα μας κατηγορήσουν όμως τότε για κρατικό παρεμβατισμό. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν ε, να επενδύσουμε περισσότερο στην συνεχή και στο περιβάλλον και να περιορίσουμε τα όσα έχουμε για τις εξωτερικές υποθέσεις. Δύο δις για τη διερμηνία. Νομίζω πως εδώ έχουμε μία κατάφορη επίθεση στην ε, πολυγλωσία και μιλάμε για θέσεις εργασίας που διακυβεύονται για ανθρώπους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ο κύριος ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστά επιλεγμένες. Θα πρέπει να ασκούμε μια στρατηγική προς τα μπροστά για τη δημιουργία νέας ανάπτυξης νέων θέσεων απασχόλησης. Και γι' αυτό λοιπόν ότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός ε, ε, θα μας δώσει τις νέες δομές. Οι συνάδελφοι που είναι υπέρ των εξοικονομήσεων στο Κοινοβούλιο να τους προτείνω να δώσουν το καλό παράδειγμα και να κάνουν αυτοί οι ίδιοι οικονομίε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δοθούν σωστές προδιαγραφέ, σαφείς προδιαγραφέ, Θέλουμε μέχρι το 2014 στον προπολογισμό να γίνουν ε, αναδιαρθρώσεις που θα μας δώσουν την ε, ικανότητα να ανταπεξέλθουμε στην κρίση. Ίσως και ο φόρος ε, επί των συναλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο για την φερεγγιότητα που θα δώσει την εγγύηση για την ε, επιστροφή των ε, πληρωμών για τις δαμόλογα. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ρούμπιξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέποντας το έγγραφο που συζητούμε, πρέπει να πω ότι δεν με εντυπωσιάζει ως έγγραφο που ε, απεικονίζει την κρίση στην Ευρώπη. Έχει ξανά τι ίδιε κατηγορίε, κάποιε παίρνουν περισσότερα χρήματα, κάποιε λιγότερε. Δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι θέλουμε να κάνουμε οικονομίε και δεν μα λέει τι θέλουμε να λύσουμε αυτόν τον προπολογισμό τώρα την περίοδο τη κρίση. Αναφέρομαι εδώ και στην κοινωνική πολιτική, επιστήμη, έρευνα, συνοχή, καθώς και τους ελέγχους και την εποπτεία οι δομέ ελέγχου και υποπτήρια στο Κοινοβούλιο εδώ Μα αναφέρουν πολύ συχνά ότι δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων ευρώ ε, βρίσκονται σε σφάλματα και χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται σωστά και χρηματοδοτούνται λιγότερο ηλεκτρικοί φορείς εδώ. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω στην Λετωνία, στη χώρα μου, στου εκλογεί μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέρντεν έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εισηγητές, και κυρίως αγαπητή συγγήτρια Φραντσέσκα Μπαλζάνη, σας ευχαριστώ όλους για την ε, σοβαρή σας εργασία. Είδαμε ότι ξεπεράσαμε ελάχιστα το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί απλώ που κρίναμε ότι είναι απαραίτητα. Δεν θέλουμε λοιπόν να ριζώνται τυφλέ περικοπέ όπω έκανε το Συμβούλιο, αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια διαρθρωμένη. Η ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεί ένα μέσο για την υλοποίηση των στόχων μα στα πλαίσια τη στρατηγική για το 2020. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε μια κρίση, θα πρέπει να δείξουμε στους συμπολίτες μας πως κάνουμε και εμείς περικοπές. Όχι όμως μειώντας προϋπολογισμούς που είναι απαραίτητοι για να χτίσουν το μέλλον τους. Θα πρέπει εμείς τις δικές μας λειτουργικές διαπάνες να τις μειώσουμε και να παγώσουμε τις αποζημιώσεις των Ευρωβουλευτών. Η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο θα είναι δύσκολη και αναμένω ε, την ημέρα που ο προπολογισμό μας θα χρησιμοποιείται από ίδιους πόρους και φοβάμαι πως ακόμα και εκτός κρίσης κάτι τέτοιο θα αργήσει να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέρντεν. Ο κύριος Σιλβέστρης θα πάρει το λόγο, επόμενος ομιλητής. Χαίρομαι, Επιτροπή Προπολογισμού, κύριε Πρόεδρε. Κατόπιν προτάσεω Επιτροπή Γεωργία, προέβλεψε αύξηση του προπολογισμού όσον αφορά το πλαίσιο που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατηγορία 2 Γεωργία και Περιβάλλον τη στιγμή της περικοπών του ΚΑΠ 110,6% σε πραγματικούς όρους. Αυτή η περικοπή δεν θα, μας, δεν θα μας οδηγήσει να πετύχουμε τους στόχους φιλόδοξης του νομοθετικού πακέτου της ΚΑΠ μετά το 2013, όπως παρουσιάστηκε εδώ και μερικές μέρες από τον Επίτροπο. Η αύξηση που ζητήσαμε στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι 200 εκατομμύρια πόρων που θα έμπαιναν για τα απορροκυπευτικά για να αντιμετωπίσουν μελλοντικέ κρίσεις όπως όλοι θυμόμαστε από το βακτηρίδιο που έπληξε πέρσι. Ελπίζω να μας δικαιώσει η ψήφο σήμερα και αναφέρομαι και σε άλλες δύο κατηγορίες, τις οποίες θέλω να υπογραμμίσω ότι μια αύξηση της κοινοτικής συνεισφοράς είναι αναγκαία. Αναφέρομαι στην πιστική βοήθεια προς τους ε, έχοντες ανάγκη, ε, χρειάζεται νομική, ε, συζήτηση νέα νομική βάση και οδηγεί στα διέξοδο στο Συμβούλιο και την τροποποίηση που ζητήσαμε επίση για την αύξηση τη δαπάνη για διαχείριση των μεταστατικών ροών, όπου εκεί η Ιταλία πλήττεται πρώτη. Ε, λόγω της γραφικής της θέσης που είναι στα άκρα της Ευρώπης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο κύριο Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα την ανταλλαγή αυτή απόψεων και μου, είναι, μου έγινε σαφές πως οι θέσεις μας εξακολουθούν να διαφέρουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάπως να τις ε, ε, προσεγγίσουμε και να πάμε στη συνδιαλλαγή ε, του Νοεμβρίου. Έχω την αίσθηση και εγώ του Ντεζαβίου γιατί νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς εξακολουθούμε να δίνουμε τη μάχη με τα ίδια στερεότυπα και με τις ίδιες προκαταλήψεις. Κάποιος είπε πως κάνετε οριζόντιες επικοπές και εσείς προκρίνετε την ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ έδειξα πολλές ε, φορές στατιστικές που αποδεικνύουν πως οι εθνικοί προϋπολογισμοί και των 27 κρατών ε, μελών αυτή τη στιγμή ε, έχουν παρουσιάσει αυξητικές τάσεις από το 2009 παρόλες τις προσπάθειες ανα, κατανομής και λιτότητας. Ε, και εμείς αντιμετωπίζουμε τους ίδιους, ε, ε, τους ίδιους περιορισμούς και ξέρουμε τι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Έχουμε το phasing in στη γεωργία, έχουμε ακόμα ανάληψη υποχρεώσεων που θα πρέπει να πληρώσουμε φέτος στα πλαίσια της έρευνας. Έχουμε τις έξτρα δαπάνες που πρικοδοτούν τα όσα έχουμε υποσχεθεί για τις αραβικές χώρες. Είμαστε λοιπόν στα στο τέλος δημοσιονομικής προοπτικές και ξέρουμε πως αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο, γίνονται πολλές πληρωμές ε, στα πλαίσια των διαστροτικών. Παρόλα αυτά, ε, στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουμε μεγαλύτερες, ε, περιορισμούς από τις εθνικού εθνικούς ε, προϋπολογισμούς, κάτι το οποίο για μένα είναι εντυπωσιακό. Καταλαβαίνετε βέβαια πως πρόκειται για μία μια παρανόηση όταν τοποθετεί κανεί τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στο 2% των εθνικών προπολογισμών. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τα έξι κράτη, και εδώ συμπεριλαμβάνω την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή αύξηση του ποσοστού στην χρηματοδότηση και μείωση της εθνικής συμμετοχής, τότε καταλαβαίνετε πως τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή οι επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, μπορεί να οδηγήσουν σε ανάπτυξη και απασχόληση και μπορεί να αποτελέσουν τη λύση του προβλήματος. Δεν πρέπει να αποτελέσουν τη ρίζα του προβλήματος, γιατί εάν ψάξει κανείς να βρει ποιο δημιούργησε το πρόβλημα, θα δει πως δεν δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο εκ μέρους του ε, Συμβουλίου στον ε, κύριο Ντομινίκ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση όσον αφορά τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό του 2012. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να σας πω ότι στο τέλος της συζήτησης αισθάνομαι ε, ότι έχω αναθαρίσει. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι πλέον κανονικά. Κατά το παρελθόν ένας μετά τον άλλον έμοιαζαν και κάθε διαδικασία προπολογισμού έμοιαζε με την άλλη. Έρχεται το Συμβούλιο με την άποψή του, αυξάνει το Κοινοβούλιο τα πάντα, το Συμβούλιο λέει καλός, αλλά δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε αυτό. Η κρίση μας ξύπνησε όλους και θα πρέπει να βλέπουμε τον προπολογισμό της Ένωσης από διαφορετική οπτική γωνία. Δίκιο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αυξάνεται ο προπολογισμό και αυξάνεται, δεν συρρυκνούται. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι η κλίμακα της ανάπτυξης. Ποιο επίπεδο ανάπτυξης και αύξησης είναι αποδεκτό από όλους. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε σε αυτό το τέλμα ε, που θα κολλούμε συζητώντας διάφορα θέματα. Θα πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες. Τι χρειάζεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι το αναπόφευκτο. Αυτό κάνουν τα κράτη-μέλη ε, κάθε χρόνο καταρτίζουν ένα προπολογισμό με περιορισμένους πόρους και θα πρέπει να επιλέξουν τις προτεραιότητές τους. Πού χρειάζονται τα χρήματα, πού πρέπει να διοχετευθούν και πρέπει να καθορίσουν ε, ποιες δαπάνες απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών τους. Σε αυτή τη φάση δεν γνωρίζουμε όμως τι πρόκειται να συμβεί Ποιο είναι το επόμενο που θα συμβεί. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι μπορεί να συμβεί σε μερικού μήνε. Εγώ ανησυχώ από την προσέγγιση του Κοινοβουλίου που θέλει να δαπανά τα αποθεματικά και να θέλει να κινητοποιήσει και το μέσο ευελιξία. Αν συμβεί κάτι μετά, τι θα γίνει, θα μα μείνουν χρήματα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτή είναι καλή πρακτική κάθε χρόνο το δημοσιονομικό Προοπτικό να αναδιαπραγματευόμαστε το πολιετές πλαίσιο δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό το πολιετέ πλαίσιο. Είχαμε καθορίσει παλιά το μέγιστο επίπεδο δαπανών, το έπαιρναν πολύ στα σοβαρά αυτό το επίπεδο όλοι και τα χρήματα υποδιαιρούνται σύμφωνα με σαφή κριτήρια και δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε κάθε χρόνο τις διαπραγματεύσει να διαλέγουμε νέα αριθμητικά στοιχεία κάθε χρόνο. Αυτό θα υπονόμευε ε, το πολιετές πλαίσιο. Θα αφαιρούσε κάθε έννοια από αυτό. Θα πρέπει να κατατήσουμε σχέδιο, ε, τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον σε αβέβαιου καιρού και θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και ισοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν μπορούμε να έχουμε μακρές, περίπλοκες ε, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και όλα τα θεσμικά όργανα να θεωρούν ότι εξυπηρετούν το λαό και ο λαός να μην ξέρει τι λένε οι θεσμοί. Τα θεσμικά όργανα χρειάζεται οι θεσμικά όργανα να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, ότι μπορούν να συμφωνήσουν εντός προκαθορισμένης χρονικής περίοδου προς όφελος όλων. Και κάτι άλλο δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Τώρα, αυτή την εποχή, μέσα στην κρίση, η συζήτηση που θα λάβει η χώρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφορά ε, το υπερβολικό χρέο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν, δηλαδή ξόδευσε πάρα πολλά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη ξόδευαν πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό μα δείχνει ένα πράγμα. Το να σπαταλάμε χρήμα δεν είναι καλή πολιτική. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν δίνει περισσότερα χρήματα για να το λύσει. Πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο αν δαπανεί περισσότερα χρήματα βοηθά την επίτευξη λύση. Ε, εδώ βρισκόμαστε τώρα εδώ έγκυται το πρόβλημα. Θα πρέπει να καθίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Το Συμβούλιο δεν αμφισβητεί τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απλώς λέμε ας καθίσουμε και ας κουβεντιάσουμε να δούμε πώς λογικά μπορούμε να παντρέψουμε τις περιορισμένους πόρους που έχουμε με τους στόχους που έχουμε να πετύχουμε. Και κάτι άλλο. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στην βοήθεια προ συγκεκριμένα κράτη-μέλη, να του δώσουμε παραπάνω χρήματα για να προωθήσουμε την οικονομία του. Να μιλήσουμε μόνο όμω το εξή. Τα χρήματα που του δίνουμε προέρχονται από το δικό του προπολογισμό καταρχά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βγάλουν, να κερδίσουν αυτό το εισόδημα, να μα το στείλουν για να το επιστρέψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στη χώρα μου, επί παραδείγματι, ε, κάθε δισεκατομμύριο που δαπανάτε για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να δαπανηθούν σε εθνικό επίπεδο, στη συγχρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιους πόρους θα κρατήσουμε στον εθνικό προπολογισμό για συγχρηματοδότηση και θα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο για δύο λεπτά στην κυρία Μπαλζάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τον Επίτροπο Λεβασδόφση και τον Υπουργό Ντομινίκη για αυτή τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και βγαίνει ένας πολύ σημαντικός παράγων. Υπάρχει μεγάλη ε, συμφωνία στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την ερμηνεία του, του προπολογισμού. Γιατί? Διότι το Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται στο να ζητά, αλλά προτείνει ε, και διάφορα επώδυνα μέτρα ε, και περικοπές στο κεφάλαιο, στην κατηγορία 4, όπως υπεθύμισε ένας συνάδελφος. Εκεί που υποφέρει, εκεί επομίστηκε περικοπές, επομίστηκε την ευθύνη να, να προτείνει περικοπές περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πρόταση που μετά από κόπους την κάναμε. Και θέλω να υπογραμμίσω όχι να χρηματοδοτήσουμε τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου, αλλά να χρηματοδοτήσουμε τι προτεραιότητε τη Ένωση. Διότι η στρατηγική του 2020 δεν είναι προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Είναι η προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να τη χρηματοδοτήσουμε, ζητώντα να χρησιμοποιήσουμε το μέσο ευελιξία για 240 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα προπολογισμό 150 δισεκατομμυρίων στο σύνολό του στα πλαίσια δημοσιονομικών προοπτικών που καθορίστηκαν το 2006, πριν από την κρίση του 2008, πριν από τη στρατηγική του 2020 και πριν από τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Σήμερα εδώ ζητάμε την χρήση του μέσου της ευελιξίας για 240 εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων εκείνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχουμε θέσει επί τραπέζης σαν ένα μέσο καταπολέμησης της κρίσης. Ελπίζω λοιπόν ότι το δικό μας κοινό όραμα στον αφάση προτεραιότητας που επανειλημμένα επεκαλέστηκε ο Υπουργό Ντομινίκ μας οδηγεί στη συνδιαλλαγή ε, σε πιο ενδελεχή καθορισμό. Είναι δύσκολο να μιλάμε για προτεραιότητες εάν δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο πολύ σημαντικό βήμα τις γραπτές αυτές προτεραιότητες να τις κάνουμε πραγματικές απτές προτεραιότητες. Το 2020 είναι αύριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για να ξεκινήσουμε να το χρηματοδοτήσουμε σαν στόχο. Και όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο οι πολίτες περιμένουν να δουν τι κάνουμε, αλλά το κάνουν και αγορές. Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά στη συνδιαλλαγή να βρούμε αυτή τη συμφωνία, μάλλον αυτή τη συμπόνια, αυτή την κατανόηση που έδειξε το Κοινοβούλιο και να κινηθούμε γρήγορα σαν αρχές του προπολογισμού σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα για δύο λεπτά το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ε, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλους τους κοιόδες εισηγητές αλλά και όλους τους ε, βουλευτές οι οποίοι επέτρεψαν να συντάξουμε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού. Ε, το έχουμε ήδη υποβάλει στο Προεδρείο και πρέπει να σας πω πως η προσπάθειά μας ήταν δύσκολη, έδωσε όμως αποτέλεσμα και επειδή ήταν πολύ ανοιχτό το Προεδρείο στις προτάσεις μας, καταφέραμε να κάνουμε αυτές τις ε, περικοπές των 74 εκατομμυρίων ευρώ ε, στον ε, προϋπολογισμό του δικού μας κοινοβουλίου στις δαπάνες μας δηλαδή. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι ε, για την διερμηνία και τη μετάφραση και τις μειώσεις και τις περικοπές εκεί. Δεν πρόκειται να οδηγήσουν με κανένα τρόπο την αρχή της πολυγλωσσίας. Η πολυγλωσία για μας είναι ιερή οι δαπάνες για τη μετάφραση και την διερμανία ε, που επιφέρουμε είναι διαθροτικές. Έτσι δηλαδή στις συνεδριάσεις επιτροπών που γινόταν παλιά Τρίτη και Τετάρτη προτείναμε να τις κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Ε, την αρχή της πολυγλωσσίας εμείς την υποστηρίζουμε από ε, πάρα πολύ παλιά και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Και για τα ταξίδια είπαμε 5% μείωση σε όλα, σε όλα τα ταξίδια. Ζητήσαμε η πρόταση να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου έτσι ώστε να έχουμε ένα απόθεμα 15% έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο αυτό τώρα για τις γενικές δαπάνες Νομίζω πως θα πρέπει το Προεδρείο να δει τι μπορεί να κάνει εκεί. Και για τη συνδιαλλαγή ζητήσαμε από το Προεδρείο και νομίζω ότι αυτό αποτελεί τμήμα του συνολικού μας συμβιβασμού να παγώσει τις δαπάνες στο τομέα αυτό. Νομίζω ότι σεβαστήκαμε τους κανόνες ε, και κάναμε κάποιες οικονομίες οι οποίες δεν ε, θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους τους οποίους έχουμε θεσπίσει που είναι η νομική, νομοθετική αριστεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προπολογισμό λιτότητας αλλά παρόλα αυτά αρκεί. Αρκεί για να σεβαστούμε τους στόχους μας. Πολύ καλά. Θα δώσω τώρα στον κύριο Μπέγκε το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς ε, να εκφράσω την ελπίδα ότι θα ακολουθηθούν οι καλές προθέσεις της Πολωνικής Προεδρίας σε έναν εντατικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προκειμένου τα ανοιχτά ζητήματα του προϋπολογισμού του 2012 να επιληθούν τον ε, Δεκέμβριο, τον Να προσθέσω επίσης ότι την περασμένη Παρασκευή και Πέμπτη στις Βρυξέλλες με την ε, συμμετοχή των ε, άλλων κοινοβουλίων χαρακτηρίστηκε από το πνεύμα ε, αμοιβαίας προσέγγισης για την εξέβρεση μιας κοινή μεθόδου προσέγγισης. Αλλά να σας πω, αξιότιμε κυρία Ντομινίκ, ότι αυτή την θετική εντύπωση κάπως την αναιρέσατε με την έκκλησή σας. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο, ως άμεσα αιρετή. δεν χρειαζόμαστε έκκληση από το Συμβούλιο για να λάβουμε τις ευθύνε μας. Ανταποκρινόμαστε στις ευθύνε μας και πολύ από το Συμβούλιο και δεν ε, ανέχομαι να μου λέει το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τους κανόνες του παιχνιδιού, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το άρθρο 120, σε ό,τι αφορά το σεβασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση 6 δισεκατομμύριων ευρώ άνω του δημοσιονομικού πλαισίου και κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων μέσων. Δεν είναι δυνατόν να α, ε, μας δίνετε τέτοιες προδιαγραφές. Ξεκινήστε κι εσείς από το του οίκου σας. Επίσης, ε, να αναφέρουμε ότι τα μέσα τα οποία διαπραγματευόμαστε, όπως το μέσο ευελιξίας ή η αναθεώρηση του πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών, αν τεθεί απαραίτητο, αποτελούν ε, τμήματα του πολιτές ε, δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να μιλάμε στα επίπεδα των υποχρεώσεων και ας μην συγκρίνουμε τα μήλα με τα χλάδια. Δεν έχουμε χρέη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφενός κατά δεύτερον ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί 37% κατά μέσο ορόνο η ευρωπαϊκή των κρατών μελών οι προπολογισμοί 62%. Άρα να μην είναι κλωτσοσκούφι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό των ε, εθνικών συμφερόντων. Αν τα καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, θα βρούμε και τη λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Πολιτισμού μέσω του κυρίου Λόκιαγκάρτ, ο οποίος θέλει να δώσει κάποιες διευκρινήσεις για τη θέση της Επιτροπής αυτής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που χρειάστηκε να λάβω το λόγο, αλλά θα τα πω στα αγγλικά πια, γιατί συνειδητοποίησα τα όσα σας είπα προηγουμένως για τη θέση της Επιτροπής Πολιτισμού ε, ε, ερμηνεύτηκε με σφαλμένο τρόπο και ίσως κάποιοι από εσά δεν κατάλαβαν γιατί ε, παραπονιέμαι για τα στοιχεία που έχουμε, ενώ αντίθετα εγώ στα Δανέζικα είπα πως με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό που έχουμε πετύχει. Αυτά για τα πρακτικά. Και πρέπει να σας πω πως πραγματικά με ανησυχούν τέτοια ίδια φαινόμενα να μη σε κατανοούν όταν μιλάς τη γλώσσα σου. Αυτά παρακαλώ για τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Λόκεγκαρτ και καταγράφουμε ε, τα λεγόμενά σας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αλλά νομίζω πως εσείς μας διαφωτίσετε για το ποια είναι η θέση σας και θα φαίνεται με σωστό τρόπο στα πρακτικά.